Right, good afternoon everybody. If you could take your seats and we'll commence the proceedings. I can see we've got a full set. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Έχουμε όλους τους εισηγητές παρόντες, παρακαλώ καθίστε. Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι μια ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τα παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους και τα μητρώα συναλλαγών. Είναι βέβαια η συγκεκριτής ο Βέρνερ Λάγκεν και το δίνω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Οι πίσω σειρέ είναι γεμάτες, ε, οι μπροστινές όχι, είναι ακόμα κενές. Θα ήθελα να κάνω κάποιες προκαταρτικές ε, παρατηρήσεις. Η ομάδα εργασία του Συμβουλίου έχει συνεδριάσει κατά επανάληψη και έχει υποβάλει κάποιες ε, προτάσεις στην Επιτροπή που δεν είναι όλες κατά την άποψή μου ενδεδειγμένες, δεν πληρούν ε, την ουσία αυτής της πρότασης, δηλαδή καλύτερη ρύθμιση της αγοράς εξωχρηματιστηριακών παραγόγων. Δεύτερον, υπάρχει η τελευταία πρόταση της 5ης Ιανουαρίου του 2011, την οποία ε, πήρε η Ουγγρική Προεδρία από τη Βελγική και την τροποποίησε ελαφρώς. Εκεί γύρεται μια γενική, ερώτηση γενικής φύσης, η οποία θα πρέπει να συζητηθεί. Κατά πόσο δηλαδή μια διεύρυνση, έτσι όπως την προτείνει η Ουγγρική Προεδρία, είναι κατά των αποφάσεων των ε, G20, των αποφάσεων της συνάντησης κορυφής και των συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με μια επέκταση της ε, πρότασης για τα εξωχρηματιστριακά παράγωγα. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει, κατά την άποψή μου, διαφάνεια και να υπάρξει και ένα αντίβαρο. Η επέκταση της πρότασης της Επιτροπής δεν είναι, ε, δεν είναι σωστό να γίνει από το Συμβούλιο. Εάν έχει αυτή την άποψη το Συμβούλιο, θα πρέπει η Επιτροπή να υποβάλει μια δική της πρόταση. Αυτό σαν αφορά το πεδίο εφαρμογής. Τρίτον, έχουμε, τρία, έχουμε αναθέσει τρία κείμενα στην επιστημονική μας υπηρεσία που ετοιμάστηκαν, ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή στην προσωρινή τους μορφή έχετε ε, τα... Ε, το έχει, τα έχει πάρει η κυρία Μπόλτς, η κυρία Μίντσου, ο κύριος Κομφά, η κυρία Σουίνμπορν και ο κύριος Γκλούτελ, οι συγητές δηλαδή και οι σκιώδεις. Αυτές οι τρεις εκθέσεις θα πρέπει να γίνουν αντικείμενα επεξεργασίας και αξιολόγησης και αφορούν ιδιαίτερα δύο από αυτές τις επιστημονικές ε, εκτιμήσεις όσον αφορά τα κατόφλια εκαθάρισης και την σύγκριση με την Αμερικανική νομοθεσία με τις ε, προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό το λόγο ε, θα ήθελα μετά από τη σημερινή συζήτηση να ολοκληρώσω την οριστική μορφή της έκθεσής μου και να τη διαβιβάσω την Τετάρτη το βράδυ στη Γραμματεία. Ε, υπάρχει εδώ, περιλαμβάνει 99 τροπολογίες και από αυτές τις τροπολογίες ένας μικρός αριθμός ε, έχουν συμπεριληφθεί από, το, από με το Συμβούλιο, από τη βουλεύση με το Συμβούλιο, ε, κάποιες από την γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ορισμένες ε, προήλθαν από την ε, πρόεδρο της Νομικής Επιτροπής. Δηλαδή προσπαθώ να καλύψω το παρόν επίπεδο των συζητήσεων και στη συνέχεια την Τετάρτη θα διαβιβαστεί η έκθεση αυτή στη Γραμματεία, ούτω ώστε να διευθούν οι προθεσμίες για την μετάφραση και την δεύτερη διαβούλευση. Ε, για σήμερα προβλέπεται η πρώτη διαβούλευση και η παρουσίαση της έκθεσης, την οποία θα κάνω προφορικά. και η δεύτερη παρουσίαση θα γίνει στις 28 Φεβρουαρίου ενώ οι προθεσμίες για τις ε, τροπολογίες είναι, η προθεσμία είναι η 15η Μαρτίου. Η διαβούλευση των συμβαστικών προτάσεων 5 Απριλίου και η ψηφοφορία στις 20 Απριλίου στην ΕΚΟΝ. Και ε, στην ε, συνέχεια θα πάνε στην Ολομέλεια του Ιωνίου. Όλα αυτά έχουν συζητηθεί με τη γραμματεία και νομίζω ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο και με την πρόταση αυτή πρόκειται να τηρήσουμε όλες τις προθέσεις ε, προθεσμίες και μπορούμε να πούμε ότι η πρόθεση του Συμβουλίου μέχρι τη συνάντηση κορυφής του, της Άνοιξης να ληφθεί μια οριστική απόφαση στο επίπεδο του Συμβουλίου, από την πλευρά της Ομάδας Εργασίας Συμβουλίου. Ναι, είναι ωραία αυτή η πρόταση, αλλά το Συμβούλιο δεν είναι δυνατόν να προγραμματίσει εκ των προτέρων κάποιες αποφάσεις που δεν έχει συζητήσει προηγουμένως με το Κοινοβούλιο. Και εγώ είμαι αποφασισμένος με τη στήριξη των συναδέλφων εδώ να εξασφαλίσω ξεκάθαρα την άποψη του Κοινοβουλίου. Τώρα, σαν αφορά τι τροπολογίε, θα ήθελα να ονομάσω εδώ τα πιο σημαντικά σημεία. Καταρχήν, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή. Αυτό το προανέφερα ήδη. Δηλαδή, ο το Συμβούλιο επιθυμεί την επέκταση του πεδίου εφαρμογή του κανονισμού για όλα τα παράγωγα. Θέλει να λάβει αυτή τη σχετική απόφαση. Αλλά υπάρχει μία μικρή ε, μειονότητα που αντιτίθεται, η οποία γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Και η αιτιολόγηση του Συμβουλίου είναι ότι ένας περιορισμός στα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα θα αφήσει κάποια κενά. Και στην έκθεσή μου εδώ ε, τονίζω ρητά ότι πρόκειται για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωνα ενώ 20% γίνονται αντικείμενα διαπραγμάτευσης στα χρηματιστήρια των παραγόγων και δεν είναι υπεύθυνα για τη χρηματοπιστωτική κρίση, ούτε μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο τη ε, πρόταση ρύθμιση εκ μέρου τη επιτροπή. Γι' αυτό πιστεύω, εάν θέλουμε να σταθμίσουμε ακριβώ τα επιχειρήματα υπέρ και κατά, μπορούμε να πούμε ότι αυτό το οποίο προτείνει η Ουγγρική Προεδρία ή το αυτό το οποίο μα ανακοίνωσε εντωμεταξύ, δεν είναι ιδιαίτερο πιστικό ότι θα πρέπει να υπάρξει δηλαδή μια γενική επέκταση τη ε, πρόταση σε όλα τα παράγωγα και όχι μόνο τα εξωχρηματιστηριακά αλλά μπορούμε να συζητήσουμε σχετικά το θέμα αυτό. Νομίζω καθοριστικό θα πρέπει να είναι το ότι η δήλωση των G20 εστιάζει στα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα όσον αφορά τη διαπραγμάτευση αλλά και την καθάριση. Ενώ οι ρυθμισμένε αγορέ υπόκεινται σε πιο αυστηρέ διατάξει. Γι' αυτό είναι απολύτω δικαιολογημένη μια τέτοια απόφαση. Η εκαθάριση στη ρυθμισμένη αγορά αυτή τη στιγμή λειτουργεί άψογα, άρα λοιπόν δεν υπάρχει ανάγκη μια επέκταση τη υποχρέωση εκαθάριση ε, σε ε, ρυθμισμένε ε, αγορέ. Και να αφορούν μόνο τα εξοχρηματιστηριακά παράγωγα. Και ένα σημαντικό θέμα είναι επίσης η εφαρμογή του Frank Act στις Ηνωμένε Πολιτείε, όπου προβλέπει ε, το, συμπερίληψη των ε, λοιπόν ε, παραγωγών στη ρύθμιση. Άρα λοιπόν θα πρέπει ε, ήδη να παρεμποδίσουμε αυτή την ε, πέκταση. Αύριο θα μιλήσω σχετικά με την Ουγγρική Προεδρία και θα πρέπει να πω ότι αν έχω τη στήριξη των συναδέλφων για την ε, διατήρηση του περιορισμού όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης, τότε το Συμβούλιο αυτή την αλλαγή όπου πραγματικά διέγραψε σε όλα τα άρθρα την διατύπωση εξωχρηματιστηριακά παράγωγα σε πάρα πολλά σημεία του κειμένου θα πρέπει να την ανακαλέσει. Δεύτερον, ένα σημαντικό θέμα είναι το ζήτημα της εξαίρεσης από τη ρύθμιση αυτή. Το άρθρο 1 γιατί εδώ έχουμε μια πληθώρα δικαιολογημένων προθέσεων σκοπών που έχουν σαν αποτέλεσμα οι διάφοροι συμμετέχοντες στην αγορά, όπως προβλέπεται από την Επιτροπή, να εξαιρεθούν γενικά. Η γενική εξαίρεση από τη ρύθμιση αυτή αντιβαίνει επίσης στις διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες και είναι προβληματική γιατί εγώ ε, θα ήθελα μάλλον να υποβάλω την προτίμηση οι εξαιρεσει να προβλέπονται, να γίνονται μέσω της, ε, ε, των, ε, μέσω της, του κέντρου Καθάρισης συμψηφισμού. Εδώ πρόκειται για τις δημόσιες τράπεζες, τράπεζες οι οποίες κάνουν διαπραγματεύσεις με παράγωγα να εξαιρούνται, να μπει δηλαδή στο πεδίο εξαίρεση από τη ρύθμιση. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ο περιορισμό, ο οποίο ε, μάλλον έχει κάποιο νόημα κάτω από συγκεκριμένε προποθέσει, δηλαδή να χορηγηθούν κάποιε εξαιρέσει για δημόσιε τράπεζε που είναι κατά 100% στην κυριότητα του κράτου, του δημοσίου. Εδώ θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Αλλά ε, και εδώ είναι δύσκολη αυτή η εξαίρεση, χωρίς εξέγερση. Και θα ήθελα εδώ να δώσουμε μία εντολή εξέτασης ε, του θέματος ε, ω αιτιολογική σκέψη. Δεύτερον, υπάρχουν συνάδελφοι που θέλουν να υπάρχει μια γενική εξαίρεση για τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Εδώ θα ήθελα να πω ότι φυσικά υπάρχουν κάποιες ε, διαφορές όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά ταμεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το σημείο αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε και θα ήθελα να προτείνω όσον αφορά αυτό το ειδικό θέμα των συνδεδετικών ταμείων ενδεχομένως να έχουμε την Συμβουλή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων. Η τρίτη επιθυμία, η τρίτη πρόταση είναι οι συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι ε, ε, έχουν δραστηριότητες στον ενεργειακό τομέα θα πρέπει να υπόκεινται σε έναν άλλο έλεγχο, όχι στον έλεγχο των παραγόγων. Αυτό το προετοιμάζει ο Επίτροπος Αρμόδιος επί της ενέργειας. Αλλά ακόμα δεν έχει ληφθεί σε αυτό το βαθμό η σχετική απόφαση. Αλλά εδώ μέσα αυτής της παρακαμπτηρίου προσπάθησα εγώ, αν θέλετε, να προσθέσω μια αιτιολογική σκέψη λέγοντας ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει στην περίπτωση αυτή όπου υπάρχει ε, μια ισότιμη ρύθμιση η οποία πληρεί τον ίδιο σκοπό να μπορεί η Επιτροπή να υποβάλει την πρόταση για εξαίρεση ενός κλάδου. Αλλά οσο έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να χωρηθεί αυτή η εξαίρεση από την Κομισιόν. Τώρα έχουμε μια ιδιαίτερη περίπτωση των ασφαλιστικών παραγόγων, όπου εδώ υπάρχουν ορισμένε μορφές παραγόγων, τα οποία ενδεχομένως όσον αφορά τα, της κατάσχεσης. Ε, ε, Όσον αφορά ε, ορισμένε ασφαλίσεις, να μην ξερούνται εν γέννη. Και Επίση έχουμε του οργανισμού για, ορισμένε κινητέ αξίε. Ε, όπου ε, είναι οργανισμοί κοινών επενδύσεων ε, σε χρεόγραφα όπου συμπεριλάμβανε μόνο σε μικρό βαθμό κάποια παράγωγα. Και εδώ θα πρέπει να δούμε σε ποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν εμπίπτουν στη ρύθμιση για τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους. Και Ε, βεβαίως υπάρχουν κάποιες ε, ιδιαίτερες ε, περιπτώσεις όπου επιχειρήσεις έχουν μικρό ποσοστό παραγόγων, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εν μέρει έχουν δραστηριότητες σε αυτή την αγορά παραγόγων. Ε, παράγω για παράδειγμα στον ασφαλιστικό τομέα. Και εδώ, στην περίπτωση αυτή, θα απαιτηθούν περαιτέρω έρευνε εκ μέρου τη Κομισιόν, αλλά δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί εξαίρεση. Με μια εξαίρεση την Τράπεζα Διακανονισμών στη Βασιλεία, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό ανταποκρίνεται και στην πρόταση η οποία υπευλήθη ήδη από το Συμβούλιο. Και στη συνέχεια μετά από αυτό το σημείο, εν σχέση με το πώς χορηγούνται οι εξαιρέσεις, πώς αντιλαμβανόμαστε δηλαδή το, τις εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογή, έχουμε το επόμενο σημείο που είναι η μη χρηματοπιστωτική αντισυμβαλόμενη, και εδώ υπάρχει μια σειρά από προβλήματα οριοθέτηση που κατά την άποψή μου έχουν σαν αποτέλεσμα η... να πρέπει να αλλάξει και η πρόταση. Στην πρόταση του Συμβουλίου είναι η διαγραφή του κατοφλίου για τις πληροφορίες. Δηλαδή μετά από ένα κατόφλι οι χρηματοπιστωτικοί αντισυμβαλόμενοι δεν έχουν την υποχρέωση αναφοράς. Στο Συμβούλιο υπάρχει μια άλλη πλειοψηφία. Ε, ε, ε, υπάρχουν ορισμένοι που λένε ότι αυτό θα δημιουργήσει ε, συγκρούσεις. Και όσον αφορά το κατόφλι μετά από το οποίο ε, πρέπει να υπάρχει υποχρέωση αναφοράς, εδώ μπορεί να γίνει μια διαγραφή εφόσον θεσπίσουμε έναν ελάχιστο κανόνα για την υποχρέωση αναφοράς, ούτως ώστε να μην είναι υποχρεωμένος ε, ο καθένας να κάνει αυτή την αναφορά σε μια μεταγενέστερη φάση, αλλά μετά την ε, καταχώρηση στο Μητρό συναλλαγή, να μπορεί να γίνει ένα έλεγχο κατά πόσο μπορούν να εκχωρηθούν ορισμένε εξαιρεσει. Αλλά ε, και με, αυτό θα πρέπει να, αυτή τη ε, διερεύνηση θα πρέπει να εκφορηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή μπορεί να συμπεριληφθεί ορισμό για το κατόφλιο, αυτό για την υποχρέωση αναφορά, αλλά από την άλλη μπορεί να θεσπιστεί αυτό ο ελάχιστο κανόνα. Δυσκολότερα είναι τα πράγματα με το κατόφλι εκαθάριση ή συμψηφισμού βάσει το οποίο θα πρέπει να γίνει η εκαθάριση των παραγόγων σε μια επιχείρηση. Με αυτό συνδέονται μια πληθώρα διαφόρων ε, προβλημάτων και εδώ θα, πρέπει, θα προσπαθήσω να το εκφράσω εξή. Το κατόφλι καθάρισης για μη χρηματοπιστωτικού αντισυμβαλόμενου είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο μέγεθος για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά. Γι' αυτό το λόγο εδώ και υπάρχουν ορισμένε προτάσεις εκ μέρους των συμμετεχόντων στην αγορά και από τι χώρε μέλη, από τι εποπτικές αρχέ των χωρών μελών, που όμω όλοι ε, δεν ε, θέλουν να προεξοφλήσουν τις αποφάσεις της ΕΣΜΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά απλώς αναφέρουν κάποια κριτήρια ε, στο παράρτημα ένα δεν θέλησα να αναφέρω όλα αυτά τα κριτήρια γιατί τα προβλήματα τυποποίησης των συμβάσεων είναι δυσεπίλητα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο ζήτημα αφορά την αξιολόγηση των διαφόρων κατηγοριών παραγόγων βάσει του κινδύνου, βάσει ε, ε, του μεγέθους κινδύνου. Δηλαδή, ε, τα παράγωγα επιτοκίων και τα, θα πρέπει να τύχουν διαφορετικής ε, αντιμετώπισης από τα CDS. Για της επιχειρήχης βάσει της επένδυσης, βάσει της αγοράς πρώτων υλών και λοιπά, βάσει διαφόρων δικτών ε, μπορούν να εξαιρούνται εδώ. Γι' αυτό η πρόταση ε, που αναφέρεται στη δεύτερη γνωμάτευση είναι να θεσπιστούν δύο κατόφλια. Ένα ε, κατόφλι το οποίο είναι ποσοτικό και ένα ποιοτικό κατόφλι ε, το ποιοτικό κατόφλι θα πρέπει να αναφέρεται στην βαρύτητα, στη σημασία της επιχείρησης στο σύνολο της αγοράς ή σε ένα τμήμα της αγοράς εξωχρηματιστηριακών παραγόγων. Κατά πόσο έχει νόημα αυτή η πρόταση ε, το αξιολογώ 0,1 μερίδιο της αγοράς σε ένα τμήμα της αγοράς ή σε μια συγκεκριμένη αγορά παραγόγων εάν ξέρουμε ότι η αγορά είναι 600 δισεκατομμύρια δολάρια. Το τμήμα αυτό των εξωχρηματιστηριακών παραγόγων εξακολουθεί να είναι αρκετά μεγάλο. Αυτό σημαίνει... Ε, βεβαίως η πρόταση αυτή δεν είναι ποσοτικοποιημένη, θα πρέπει να γίνει αυτό βάσει άλλης εξέτασης. Τώρα, όσον αφορά την ανάγκη προσανατολισμού στο μέγεθος ισολογισμού, στην, ε, στο κίνδυνο, στο πιστοτικό κίνδυνο σε κάποιους άλλους παράγοντας η πρόταση λέει ότι αν ε, συντρέχει ένας αυτός παράγοντας θα πρέπει να γίνεται μια εκαθάριση και αυτό είναι το πιο δύσκολο έργο της ΕΣΜΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή να ορίσει ακριβώς αυτό το κατόφλι και να μπορεί επίσης να το επαληθεύσει, ε, κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει μέχρι το 2012. Και θα πρέπει να πω ότι αυτό είναι το πιο βασικό από την πλευρά των επιχειρηματιών, δηλαδή το που θα οριστεί ακριβώ αυτό το κατόφλι για το συμβισμό την εκαθάριση. Από την άλλη, είναι δυνατόν, ε, θα πρέπει να γίνει μια ε, τυποποίηση των συμβάσεων ή δυνατόν ε, η μεγαλύτερη δυνατή όσον αφορά τον κίνδυνο του αντισυμβαλόμενου. Τώρα, ε, σε μια περαιτέρω φάση ΕΣΜΑ θα πρέπει να εξετάζει κατά πόσο θα πρέπει να θεσπιστεί μια, ένας ελάχιστος κανόνας ε, για το ελάχιστο όριο για την υποχρέωση αναφοράς. Βάσει της πρότασης ε, στους μη χρηματοπιστωτικούς ε, αντισυμβαλόμενους η υποχρέωση για την καθάριση ή το συμψηφισμό στοιχίζει χρήματα. Αυτό είναι ξεκάθαρο γιατί οι συναλλαγές αυτές υπολογίζονται εφόσον ξεπεραστεί το κατόφλι της εκαθάρισης. Από την άλλη δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι οι επιχειρήσεις ε, εν γέννη δεν ε, έχουν καθόλου κινδύνους μέσω των παραγόγων. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει βάσει κανόνων μια εξέταση. Ένα τρίτο σημείο είναι πότε ισχύει η υποχρέωση αναφοράς καθάρισης. Ε, άπαξ εφόσον ξεπεραστεί το κατόφλι αυτό ή αργότερα σε μια μεταγενέστερη φάση. Η πρότασή μου είναι ότι η υποχρέωση, αναφοράς, η υποχρέωση καθάρισης θα πρέπει να ισχύει εφόσον επί 90 μέρες έχει ξεπεραστεί το κατόφλι αυτό της εκαθάρισης, το οποίο όμως προηγουμένως θα πρέπει να έχει οριστεί. Και στη συνέχεια επιχειρήσεις θα πρέπει να προσπαθήσουν να τα απεξέλθουν στα καθήκοντά τους. Στις νέες συμβάσεις αυτό ισχύει ευθύς εξ αρχής για τις παλαιές συμβάσεις, για το backloading, ε, σκέφτομαι που σας ανέφερα και θα πρέπει να πω επιπλέον ότι σε αυτό το backloading, δηλαδή οι επιπλέον, ε, για τις επιπλέον συμβάσεις ισχύουν μόνο εκείνες ε, οι συμβάσεις που την ημέρα της εκαθάρισης η σύμβαση ισχύει για δύο ακόμα χρόνια. νομίζω ότι αν μία μέρα μετά την υπέρβαση του κατοφλίου εκαθάρισης, όπως λέει η Κομισιόν, ισχύει η υποχρέωση εκαθάρισης για, όλες, για όλα τα παράγωγα, ε, τότε θα επιβαρυνθεί η κεφαλαϊκή ε, βάση όλων των επιχειρήσεων και δεν είναι δυνατόν με τον τρόπο αυτό να ταποκριθούμε στην ε, ανάγκη, στο σκοπό ελαχιστοποίηση των ε, κινδύνων. Εάν θέλουμε λοιπόν να ταποκριθούμε σε αυτή την υποχρέωση καθάριση και να δούμε ε, σε σχέση με τις ευκταίε εξαιρέσει από το πεδίο εφαρμογή που θα πρέπει να χορηγηθούν, προσεγγίζουμε κάπως το σωστό μοντέλο. Εγώ θα έλεγα, θα πρότεινα οι θηγατρικές εταιρείες, ε, αν έχουν ενωπημένους λογαριασμούς, αν έχουν μια κυριότητα της τάξης του 50%, τότε ε, θα πρέπει ε, στις συναλλαγές τους με τις τρεις χώρες να μην έχουν μια υποχρέωση καθάρισης, γιατί στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση εκαθάρισης ε, για επιχειρήσεις που έχουν μια διεθνή δραστηριότητα και που δεσμεύονται με παράγωγα έχει νόημα εφόσον η επιχείρηση που έχει μία έδρα στην Ευρώπη ε, διεκπεραιώνει μόνο το ένα τμήμα των συναλλαγών που αφορά την Ευρώπη ενώ το άλλο κομμάτι των ε, παραγόγων ε, χάνεται. Τώρα, όσον αφορά τις άδειες για τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους, εδώ έχω τις προτάσεις του συναδέλφου Σκίνερ, δεν ε, παρίσταται εδώ, τις έχω συμπεριλάβει, λέει ο συνάδελφος, ε, αναφέρεται στα όργανα τα οποία έχει προτείνει η Επιτροπή και τα οποία τελικά συνιστούν μια επιπλέον επιβάρηση και παρεμποδίζουν μια αποτελεσματική ρύθμιση. Ε, θεωρώ ότι οι χώρες οι οποίες ε, φύγονται δευτερογενώς μόνο από τη ρύθμιση αυτή ε, dass die, die Clearingpflicht äh, äh, Εκεί, εδώ η υποχρέωση εκαθάρισης δεν θα πρέπει να παρεμποδίζονται από γραφειοκρατικές διαδικασίες όπως προβλέπεται από την γνωμοδότηση του συναδέλφου όπου στο τέλος ε, θα πρέπει να συμφωνήσουν τουλάχιστον 50 άτομα για μια κοινή γνωμοδότηση. Γι' αυτό ε, συμπεριέλαβα εδώ την ε, πρόταση του συναδέλφου Σκίνερ να καταρριχθούν αυτά τα συλλογικά σώματα, αλλά η ΕΣΜΑ να διαβουλεύεται το Ευρωπαϊκό Σύστημα των Κεντρικών Τραπεζών και να διαβουλεύεται με τους συμμετέχοντες στην αγορά πριν από την υπέρβαση του κατοφλίου αυτού και θα πρέπει επίσης να έρθει συνεννόηση με τις εποπτικές αρχές των χωρών που ενδιαφέρονται εδώ ε, ούτως ώστε να καταλήγουν σε μια κοινή γνωμοδότηση. Και εδώ είναι σημαντικό αυτές οι προτάσεις να προτείνονται επίση και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να γίνονται σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική ε, Τράπεζα. Η χορήγηση αδειών δεν θα, γίνεται, δεν πρέπει να γίνεται μέσω ενός οργάνου, συλλογικού οργάνου, το οποίο ευθύνη δεν ορίζεται επακριβώ. Γι' αυτό η χορήγηση άδεια για ένα κεντρικό αντισυμβαλόμενο θα, θα πρέπει να γίνεται σε μία ε, δεν θα πρέπει να γίνεται σε όλες τις χώρες μέλη, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίζεται από την ΕΣΜΑ να είναι απολύτως ξεκάθαρες οι προϋποθέσεις, να μην ε, γίνεται δηλαδή αυτό το οποίο είχε συμβεί στην ε, Ιρλανδία. Εδώ θα ήθελα να πω ότι περιλαμβάνω τις απόψεις του συναδέλφου κυρίου Σκίνερ. Όσον αφορά τώρα την ενίσχυση των χωρών μελών για την έγκριση των κεντρικών αντισυμβαλόμενων από τρίτες χώρες. Εδώ η πρόταση της Επιτροπής κατά την άποψή μου είναι υπερβολικά μετριοπαθής και θα πρέπει εδώ να δημιουργήσουμε ισότιμους όρους ε, και θα ήθελα αυτό να το τονίσω ρητά. Ε, σε αυτό το σημείο προτείνεται η έγκριση από κεντρικούς αντισυμβαλόμενους τρίτων χωρών να ρυθμίζεται ακριβώς όπως οι άδειε για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με μια προσθήκη, η Κομισιόν έχει μια άδεια χορήγηση εξαιρέσεων, δηλαδή μπορεί να χορηγήσει μια άδεια για ένα κεντρικό αντισυμβαλόμενο εφόσον υπάρχει διμερή συμφωνία με το εν λόγω τρίτο κράτος όσον αφορά την ισότιμη άσκηση, διενέργηση ελέγχου. Και εδώ βλέπετε ότι έχω συμπεριλάβει την πρόταση Κομισιόν. Τώρα έχουμε την επόμενη, το επόμενο σημείο που αφορά τη διαλειτουργικότητα. Εδώ η Επιτροπή ήταν ιδιαίτερα συγκρατημένη όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον ισχύει για όλα τα παράγω και επεκταθεί σε όλους τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους, θα ε, προσδώσει εντελώς νέες ε, διαστάσεις. Γι' αυτό η Κομισιόν έκανε κάποιες άλλες προτάσεις για τη διαλειτουργικότητα. Εγώ θα πρότεινα να διαγραφούν εν γέννη αυτές οι διατάξεις και να επιφορτήσουμε την Κομισιόν με την εντολή αργότερα να επεξαρτηθεί το ζήτημα της λειτουργικότητας στη βάση μιας πλήρους διαφάνειας των στοιχείων. Γι' αυτό όλο το κεφάλαιο 5 έχει διαγραφεί εκ μέρους μου γιατί ε, προποθέτει μια προηγούμενη εξέταση η οποία όμως συνδέεται με μια αύξηση συστημικών κινδύνων. Και ε, στη συνέχεια έχουμε μια πληθώρα καθηκόντων της ΕΣΜΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το στόχο της συμμετοχής των συμμετεχόντων στην αγορά, στην ε, προετοιμασία ε, του Ευρωπαϊκού Συστήματος των Κεντρικών Τραπεζών. Και αυτά τα ζητήματα που αφορούν στην τυποποίηση θα πρέπει να ολοκληρωθούν το πρώτο ίμιση του 2012 στα μέσα του 2012 θα έχουμε ε, τις προτάσεις της ΕΣΜΑ και της ε, Κομισιόν και ε, κάτι που είναι εξαιρετικά πολύπλοκο βεβαίως, αλλά νομίζω ότι βάσει της ρύθμισης στις ΗΠΑ και των δικών μας ε, προβληματισμών μπορούμε να αξιοποιήσουμε το χρόνο μέχρι τώρα. Όσον αφορά τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους, εδώ πρόκειται και ε, συνδέονται με το ζήτημα των ε, κανόνων για την εσωτερική εποπτεία, για την διακυβέρνηση, τους εσωτερικούς ελέγχους, κινδύνων και εδώ θα ήθελα να προτείνω η Προεδρία στην ομάδα διερεύνησης του κινδύνου ε, να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Εδώ έχουμε κάνει κάποιες δικαιολογημένες παρατηρήσεις σε σχέση με τη ρύθμιση της αφερεγγυότητας για τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους. Εδώ νομίζω είναι πολύ καλή η Επιτροπή της Κομισιόν. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε, έτσι τουλάχιστον η πρόταση της Επιτροπής, εάν ε, σε, ένα, σε μια εκαθάριση ε, χρεοκοπήσει ο μεγαλύτερος πελάτης και συνέχεια ο δεύτερος μεγαλύτερος και ο τρίτος μεγαλύτερος, θα πρέπει να υπάρχει, ε, θα πρέπει να εξασφαλίσει την κεφαλαϊκή επάρκεια και θα υπάρχει ένας επαρκής διαχωρισμός γιατί ξέρετε ότι διάφορες χώρες μέλη υπάρχουν διάφορες ε, ε ρυθμίσεις ε, για τα θέματα φεργιώτες. Γι' αυτό αυτή η παράγραφος είναι ιδιαίτερα σημαντική. Τώρα, όσον αφορά το μητρό συναλλαγών ε, για κάθε κατηγορία παραγόγων και για κάθε χώρα μέλος, ε, πόσες θα πρέπει να εγκριθούν, πόσες άδειες θα πρέπει να χορηγηθούν. Έχουμε δύο σημαντικά μητρώα καταγραφής, τα οποία υπάρχουν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις Ηνωμένε Πολιτείε, για παράδειγμα, που καλύπτουν 80% των παραγόντων των έξι μεγαλύτερων συμμεταχόντων στην αγορά, που έχουν ένα τεράστιο κομμάτι της αγοράς σε παράγωγα και όπου καταγράφονται όλα αυτά, καταχωρούνται σε εθελοντική βάση. Το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να πετύχουμε στον τομέα αυτό να δώσουμε μία άδεια για τα μητρώα συναλλαγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξασφαλίζοντας την ε, πρόσβαση ε, σε αυτά τα μητρώα καταγραφή συναλλαγών στις τρίτες χώρες. Και αυτό το λέω γιατί έσμασε μια από τις ακροάσεις της, αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην ομάδα εργασία του Συμβουλίου είπε ότι δεν είναι σε θέση, δεν θεωρεί ότι είναι σε θέση με το ε, περιορισμένο της προσωπικό και ενόψη τη πληθώρας των καθηκόντων που έχει να μπορεί αυτοτελώς άμεσα και αποτελεσματικά να ε, δημιουργήσει αυτό το Μητρό καταγραφή Συναλλαγών. Ε, θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια ρύθμιση σε σχέση με τα μητρώα καταχρήση συναλλαγών των τρίτων χωρών. Και εδώ η πρόταση της Επιτροπής συνολικά είναι θετική. Και θα ήθελα όσον αφορά αυτά τα σημεία μετά τις ε, διαβουλεύσεις σήμερα και μέχρι Τετάρτη το βράδυ να τα οριστικοποιήσω και θα ήθελα επίσης να σε ευχαριστήσω θερμά, να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους, τους σκιώδεις, και τις ε, αρχές των χωρών μελών, αλλά και όλου τους συμμετέχοντες στην αγορά που μπόρεσαν ε, πράγματι να μας βοηθήσουν. Την τελευταία απόφαση βεβαίως την έχουμε εμείς, ο κάθε συνάδελφος, ο οποίος μπορεί να υποβάλει τροπολογίες, ο συνήθως, και ε, δεν θα πρέπει να απομακρυνθούμε από την πρόθεση του Συμβουλίου και της Ουγγρικής Προεδρίας να υποβληθεί ένα κείμενο μέχρι τις 20 Μαρτίου. Εμείς θέλουμε στις 20 Απριλίου να υπάρχει η δική μας ε, γνωμοδότηση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αποβάλουμε μια τροποποιημένη ε, πρόταση μέχρι τα μέσα του χρόνου. Μια τελευταία παρατήρηση. Θεωρώ ότι είναι αναγκαίο στο πλαίσιο αυτό να συζητήσουμε και για το προσωπικό και για την ιεράρχηση των αρχών, ε, των ρυθμιστικών αρχών. Αυτό το λέω γιατί σήμερα ακούσαμε τους υποψήφιους ε, ε προέδρους τριών εποπτικών αρχών, ρυθμιστικών αρχών, εποπτικών αρχών και σχημάτισα την ε, άποψη ότι δεν υπάρχει βούληση να πρικοδοτηθούν αυτά τα θεσμικά εποπτικά όργανα επαρκώς και σε συμφωνία με το πνεύμα του Κοινοβουλίου. Ε, σας ευχαριστώ και Συγγνώμη που ε, παρέθεσα τόσο πολλές τεχνικές λεπτομέρειες. Να περάσουμε στους κοιόδης. Θέλω να πω στον εισηγητή ότι πολλές φορές έχουμε συζητήσεις με την Προεδρία όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα Δεν θέλουμε να μας πιέσει κανείς, ιδιαίτερα όσον αφορά την ολοκλήρωση και τη διαφάνεια της εργασίας μας. Για τη σοσιαλιστική ομάδα. Ο κύριος Ντομένετσι. Ε, η δική μου παρέμβαση θα είναι σύντομη. Γιατί πιστεύω ότι μετά την ε, ευρύτατη εισήγηση του κυρίου Λάγκεν, χρειάζεται τώρα να εμβαθύνουμε στις ε, μεμονωμένες πτυχές και να συνεργαστούμε καταρχήν για να τηρήσουμε τα χρονικά περιθώρια που έχουμε στη διάθεσή μας. Να κάνω μόνο κάποιες παρατηρήσεις. Η πρώτη αφορά το τελευταίο τμήμα της παρέμβασης του Λάγκεν, καθώς και τα όσα είπε η Πρόεδρος. Πιστεύω πως πρέπει όντως να κάνουμε καλή δουλειά, αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται να σεβαστούμε το χρονοδιάγραμμα. Και γι' αυτό νομίζω πως θα ήταν χρήσιμο να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων για την οργάνωση της δουλειάς μας ως Επιτροπή εδώ, προβλέποντας, και είναι μια πρόταση που υποβάλλω, τη δυνατότητα για μια δημόσια ακρόαση που θα μπορούσε να διοργανωθεί πριν από την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή των ε, τροπολογιών αλλά για να έχουμε μία άμεση επαφή με τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς που θα αντιπροσωπεύονται εδώ με ισόρροπο τρόπο. Τώρα, κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτη, εγώ συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με την ε, έκθεση του κυρίου Λάγκη. Την πρώτη παρατήρηση που έχω να κάνω αφορά αυτό το σημείο που αφορά την, την κατάργηση της ε, αναφοράς στα OTC, over the counter. Νομίζω και εγώ ότι το επίκεντρο της προσοχής μας θα πρέπει να είναι ακριβώς τα over the counter. Γιατί γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε η έκθεση πρωτοβουλίας και στη συνέχεια ο κανονισμός και θα τα πω τώρα έτσι σύντομα. Όσον αφορά τις εξαιρέσεις, συμφωνώ για το γεγονός ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε εξαιρέσεις ε, γενικευμένες και προσωπικά ε, φρονώ ότι σε αυτό το σημείο εφόσον η διχωριστική γραμμή που θα πρέπει να τραβήξουμε είναι πολύ περίπλοκη, θα ήταν σκόπιμο να δοθούν κατευθύνσεις επί των οποίων στη συνέχεια θα είναι δυνατόν να γίνει τεχνική εφαρμογή. Για τα μη χρηματοπιστωτικά αντισταθμίσματα, νομίζω πως θα πρέπει να δουλέψουμε για αυτό το κριτήριο το ποιοτικό και το ποσοτικό για το οποίο έκανε λόγο ο Λάγκεν. Αλλά ταυτόχρονα να αφήσουμε το κατόφλι συμψηφισμού, ιδιαίτερα όσον αφορά την τάξη μεγέθους, γιατί είναι ένα από τα πιο λεπτά ζητήματα αυτό. Τώρα, για την χορήγηση αδείας για τα κεντρικά, τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους, ο Λάγκεν είπε ότι συμφωνεί με το Σκίνερ και εγώ νομίζω πως είναι σωστό να ξεπεράσουμε ή, εν πάση περιπτώσει, να απλοποιήσουμε τη σημερινή δομή που φαίνεται να είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Νομίζω ότι ως προς αυτό είναι απαραίτητο να υπάρξει στενή συνεργασία ανάμεσα στην ΕΑΚΑ και τις εθνικές αρχές εποπτείας. Τώρα για τη διαλειτουργικότητα δεν νομίζω ότι μπορούμε ακόμα να κάνουμε ε, τις σωστές ε, εκτιμήσεις όσον αφορά την κατάργηση του τίτλου 5 και τέλος ε, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο και εδώ αναφέρομαι και στην ε, ακρόαση που είχαμε σήμερα το πρωί, να επιμείνουμε ως Κοινοβούλιο και ως Κομισιόν ώστε να υπάρχουν όλα τα μέσα στη διάθεση της αρμόδιας αρχής ώστε να μπορεί να υλοποιήσει την δραστηριότητα που όσον αφορά την καταγραφή και τον έλεγχο των συναλλαγών που έχουν ιδιάζοντα τεχνικό χαρακτήρα. Μια τελευταία παρατήρηση γιατί Φυσικά ο δικός μας χρόνος είναι ο χρόνος της συζήτησης και της δημοκρατίας, αλλά ο κόσμος εντωμεταξύ κινείται. Πιστεύω ότι θα ήταν απαραίτητο να καταλάβουμε τι συνέβη αυτούς τους μήνες και τι συμβαίνει ακόμα και τώρα. Εγώ θα ήθελα να θυμίσω και να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα σημείο όλος ιδιαίτερο για να δούμε κατά πόσο είναι σκόπιμο να βάλουμε στο εσωτερικό του κανονισμού μια κάποια αναφορά ή εν πάση περιπτώσει να ε, συνοδέψουμε τη γνωμοδότησή μας με συγκεκριμένες υποδείξεις και αναφέρομαι ιδιαίτερα στο θέμα των παραγόγων στον τομέα των γεωργικών και αγαθών και των τροφίμων, το commodities market και πιο συγκεκριμένα στο food και agricultural market, όπου διαπιστώσαμε τελευταία περίοδο μια τάση ιδιαίτερα ανησυχητική για φαινόμενα κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Και διρωτάμε σε αυτή την περίπτωση μήπως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτή την πτυχή Όσον αφορά τον κανονισμό μας, ευχαριστώ τον κύριο Λάγκε για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα και εύχομαι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας και να ολοκληρώσουμε εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι σκιώδης για την ομάδα ALDE και θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια εδώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την εξήγηση των όσων περιλαμβάνονται στην έκθεσή του. Νομίζω πως έχει κάποιες ενδιαφέρουσες ιδέες που μπορεί όντως να λειτουργήσουν. Θα πρέπει να πω ότι κάποιες πτυχές της του καθολικού πεδίου εφαρμογή ε, με έβαλαν σε πειρασμό, αν και εγώ θεωρώ πως θα πρέπει περισσότερο να τονίσουμε το τμήμα καταγραφής όλων αυτών των στοιχείων, ώστε να έχουμε δηλαδή όσο γίνεται περισσότερα στοιχεία διαθέσιμα. Και περιμένω να δω ακριβώς τι θα προτείνετε, και είπατε ε, ότι στο πλαίσιο των εξαιρέσεων και τα λοιπά θα γίνονται εξαιρέσεις μόνο όταν υπάρχουν ε, αντιστοιχίες. Και ίσως αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στις συναλλαγές, όταν υπάρχει δηλαδή κάποια αντιστοιχία στον τρόπο με τον οποίο συμψηφίζονται οι συναλλαγές αυτές. Αυτό είναι ικανοποιητικό. Αλλά υπάρχει και η πλευρά του Μητρώου και της καταγραφής. Επίσης με ανησυχεί κάπως το πώς θα συνδέσουμε τα όσα κάνουμε εδώ με την οδηγία περί κεφαλαικών απαιτήσεων, διότι φυσικά θα υπάρξουν επιπτώσεις και εκεί. Και είναι κάπως ατυχές ότι δεν το κάνουμε αυτό συν τα σχετικά στοιχεία του MIFID και τη CRD4 ταυτόχρονα. Και δεν ξέρω πώς θα τα συντονίσουμε όλα αυτά, γιατί κατά κάποιο τρόπο εμείς εδώ σε αυτό το κείμενο προσπαθούμε να διορθώσουμε κάτι χωρίς να ξέρουμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις σε άλλα κείμενα που με τη σειρά τους θα μπορούσαν να αλλάξουν τη γνώμη μας για τις εξαιρεσει. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε πώς το σκέφτεται ακριβώς η Κομισιόν. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε ακριβώς. Ίσως να πρέπει να σκεφτούμε και πράξη κατεξοδότηση αν αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να λειτουργήσουμε επίσης. Ε, το θέμα των εξαιρέσεων για τις συντάξεις ε, ήταν ένα ελκυστικό επιχείρημα, γιατί, αλλά βέβαια και εκεί εξαρτάται πώς θα χειριστούμε τις ε, παρενέργειες σε άλλα προϊόντα. Και εκεί αν βρούμε μια λύση ε, θα πρέπει να εξετάσουμε τις επιπτώσεις στο CRD4 και αλλού. Ίσως να μην χρειάζεται να εξαιρεθούν αν βρούμε τη σωστή ε, μεταχείριση. Γιατί όντως η σύνταξη, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ γιατί η σύνταξη του απλού ανθρώπου είναι αυτή που θα κινδυνεύσει. Τώρα για τα κατόφλια είναι πολύ σημαντικό όταν ε, ξεπερνάτε ένα κατόφλι να μην διατηρείται η αξία Μάλλον να μην αλλάζει διαρκώ η αξία του παραγόγου και να έχουμε ένα εφέ γιο-γιο ότι τώρα είσαι πάνω, τώρα είσαι κάτω, τώρα είσαι πάνω και ξανά κάτω και ούτω καθεξής. Να μην αρχίζει δηλαδή η εκ νέου υπολογισμός της αξίας από τη στιγμή που υπερβαίνει κανείς για λίγο το κατόφλι. Τώρα, το backloading. Ενδιαφέρουσα ιδέα. Υπάρχει βέβαια το νομικό ζήτημα για το κατά πόσο έχει δοθεί κατάλληλη ενημέρωση για την ε, πιθανότητα υπάρχ, ε, του να υπάρξει ένας αναδρομικός νόμος, μια, ένας νόμος με αναδρομική ισχύ και επίσης δεν ξέρω κατά πόσο όλα αυτά μπορούμε να τα καθορίσουμε εφόσον η ΕΕΚΑ θα πρέπει να προχωρήσει σε μια διαδικασία όπου θα επιλέξει διάφορες κλάσεις για συμψηφισμό. Οι, κεντρικοί συμβαλόμενοι θα τα οργανώσουν όλα αυτά από κοινού και ξαφνικά ανακαλύπτουν ότι ισχύουν αναδρομικοί κανόνες. Ε, μπορεί αυτό να οριστεί από να, να, να είναι καθοριστικό μάλλον το ημερομηνίες ισχύως Αλλά και εδώ ανησυχώ πως τελικά καλύψουμε πράγματα τα οποία δεν αξίζει τον κόπο να καλύψουμε. Γιατί μιλάμε βασικά για στοιχεία τα οποία σχετίζονται με υποδομές και για πράγματα τα οποία είναι σχετικά ασφαλή. Και πιθανότατα φτιάχνουμε ένα σωρό δουλειά για σχετικά ισχνά αποτελέσματα. Με ανησυχεί λοιπόν όλο το θέμα αυτό του backloading, της αναδρομικής ισχύω ε, νομοθεσιών, αν και ξέρω πού βασίζονται όλα αυτά. Ας πούμε να έχουμε την αναδρομική ισχύ για τα μητρώα, ώστε να έχουμε σε κάποια στιγμή τα στοιχεία στη διάθεσή μας. Εκεί αξίζει τον κόπο. Και έτσι νομίζω ότι καλύπτονται οι περισσότεροι σε πτυχές κινδύνου. Όμως ίσως και αυτό να μην είναι τελικά ζήτημα, γιατί γιατί μπορεί τελικά η κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι να μπορέσουν να αντιπαρέλθουν όλα αυτά τα προβλήματα λόγω του ότι θα μπορέσουν να προλάβουν τις, τις ρήτρε για τα τοξικά παράγωγα. Τώρα, για τις εξαιρέσεις ε, τις εταιρικές. Αυτές θα μπορούσαν να ελεγχθούν μέσω των ε, λογιστικών ελέγχων. Αυτό μπορεί να σταθεί όταν έτσι εξασφαλίζεται πως η χρήση των παραγωγών είναι κάτι το οποίο γίνεται μόνο από τις αρμόδιες επιχειρήσεις και όχι κάτι το οποίο ήταν γενικά γενικευμένο, δηλαδή σαν να γινόταν ας πούμε, ένα παραχρηματιστήριο, όπως έκανε ένας ε, δια, περίφημος ε, αυτοκινητοβιομήχανος και προχώρησε στο short selling. Ναι, τα ξέρουμε τα καμώματα της Porsche, όλοι μην στεναχωριέστε. Ε, Επίση έχουμε... Κάπως συμφωνούμε σε σχέση με τα όσα είπε ο Ντομένιτς ε, για τις ροές ε, δεδομένων, γιατί όλα αυτά καταλήγουν στις τράπεζες επενδύσεων. Εγώ δεν έχω τόσο απόλυτη άποψη για το πού θα συγκεντρώνονται όλα αυτά, <clears throat> αλλά είναι σημαντικό να καταλήξουμε. Αυτά λοιπόν είναι τα σχολεία μου για τώρα. Έχω και άλλα, αλλά έχουμε και άλλους ομιλητές. Ε, θα ξεπεράσουμε λίγο το χρόνο μας. Θα μπούμε και στον χρόνο της ψηφοφορίας, γιατί έχουμε μια ώρα για την ψηφοφορία προβλέψη, αλλά δεν νομίζω πως θα χρειαστούμε μια ώρα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο αυτό για να συνεχίσουμε τη συζήτηση για τα παράγωγα. Επόμενο και είναι τώρα για τους πράσινους, ο Πασκάλ. Ναι. Είναι δύσκολο να συζητήσουμε για μια έκθεση ενώ δεν την έχουμε μπροστά μας. Αλλά θα βασιστώ στην πάρα πάρα πολύ λεπτομερή σας παρουσίαση. Αλλά όπως ξέρετε με τη μετάφραση πολλές φορές δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έχω λοιπόν κάποιες ερωτήσεις. Είπατε ότι λαμβάνετε υπόψη σας και συμφωνείτε με τις τροπολογίες του Σκίνερ όσον αφορά την κατάργηση των συλλογικών αυτών ε, οργάνων, σωμάτων. Ποιος τελικά όμως δίνει την άδεια και ποιος αναλαμβάνει τη ρύθμιση, την καθημερινή, πώς γίνεται η εποπτεία, ο έλεγχος, από τη στιγμή που οι διαφορετικοί κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι δεν χρησιμοποιούν την, τον ανταγωνισμό στα μοντέλα κινδύνου τους. Ένα από τα πιο σημαντικά διακυβεύματα αυτής της, εποπτή, εποπτείας είναι να αποφύγουμε η εκαθάριση να γίνεται με διαφορετικά μοντέλα κινδύνου. Και αυτό ήταν ενδιαφέρον όταν υπήρχαν εφωτά συλλογικά σώματα, διότι γινόταν ένας ανταγωνισμός ε, και μια εποπτεία συλλογική σε όλους αυτούς τους τόπους όπου γίνεται ο συμψηφισμός. Για να υπάρχει ο έλεγχος και του συστημικού κινδύνου και του κινδύνου ε, αυτό που επίσης είναι πολύ σημαντικό είναι το θέμα της ρευστότητας της κεντρικής τράπεζας. Δεν κατάλαβα τι είπατε ακριβώς, ε, πού θέλετε δηλαδή να φτάσουμε. Συμφωνείτε με τις προτάσεις της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Την συμπεριλαμβάνετε και αυτήν στην εποπτεία. Και, εν πάση περιπτώσει, τι άδεια δίνεται όσον αφορά τη ρευστότητα της Κεντρικής Τράπεζας. Ποιο είναι το επίπεδο. Τρίτη ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω το φάσμα σε σχέση με την αμερικανική ρύθμιση. Ξέρω ότι υπάρχει το CTC και FTC. Δεν έχουν πάρει ακόμα απόφαση οι Αμερικανοί όσον αφορά τη δική τους κανονιστική ρύθμιση. Η ACC, η FTC είναι αυτή που θα παίζει αυτό το ρόλο. Όλες οι συναλλαγές θα λαμβάνονται υπόψη ή μόνο στις Ηνωμένε Πολιτείες και όσον αφορά τις συναλλαγές παραγόγων θα ελέγχονται αυτές και από τις ευρωπαϊκές και από τις αμερικανικές αρχές όταν λαμβάνουν χώρες στην Αμερική. Δεν ξέρω τι απόφαση έχει ληφθεί και δεν ξέρω εάν έχετε ξεκινήσει συζητήσεις με την ACC και την FTC. Θα ήταν κρίμα ο Ευρωπαίος νομοθέτης να αναγκαστεί να δεχτεί κανόνες που καθορίζονται από τους Αμερικανούς και να αναγκαστούμε εμείς απλώς να τους δεχτούμε και να προσαρμοζούμε. Δεν θέλω να μου πείτε ποια είναι η δική σας θέση και αν συνεργάζεστε και πώς με τους Αμερικανούς. Τέλος, συμφωνώ με τον Λεωνάρδο και την Σάρον όσον αφορά τις πρώτες ύλες, τα commodities. Το θέμα αυτό με βρίσκει σύμφωνο. Πρώτον, επειδή είναι πολύ σημαντικό το θέμα των πρώτων είναι ένα θέμα που έχει αναλάβει σαν προτεραιότητα η Προεδρία η Γαλλική του G20. Μας αφορά ιδιαίτερα το θέμα των γεωργικών πρώτων Και δεύτερον, για το interoperability, τη διαλειτουργικότητα. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε να αναβληθεί το σημείο αυτό για αργότερα. Ευχαριστώ. Okay. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τις πολύ πλήρεις ε, λεπτομέρειες που μας παρουσίασε. Κατάλαβα πολύ καλά που θέλει να πάει, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν τέσσερις πτυχές που μας ανησυχούν παρόλα αυτά. Το backloading, το θέμα των ε, συντάξεων, των συναλλαγματικών ισοτιμιών, και καταρχήν θα ήθελα να πω αυτό που αρχικά μας ε, παρουσίασε ο κύριος Λάγκεν. Μιλάμε μόνο για τα OTC ή για όλα τα παράγω. Η φιλοδοξία του G20 είναι να μειωθεί ο κίνδυνος και όσον αφορά τα προϊόντα αυτά και όσον αφορά τον συμπληφισμό. Τι θα παραμείνει όμως στον χώρο του OTC και τι ακριβώς θα ρυθμίσουμε και αν οι κανόνες αυτοί ισχύουν μόνο για το OTC, ένα μεγάλο τμήμα των συναλλαγών που λαμβάνουν χώρα σήμερα στο χώρο των OTC δεν συμπεριλαμβάνουν τα λεγόμενα OTF Θα συνεχίσουν λοιπόν να βγαίνουν από το χώρο των OTC κάποια προϊόντα, κάποια παράγωγα, γιατί αλλιώς θα παραμείνει ένας ελάχιστος αριθμός συναλλαγών σε αυτό το χώρο. Άρα θα ρυθμίσουμε έναν ελάχιστο ε, αριθμό συναλλαγών. Μήπως λοιπόν πρέπει να δούμε ακριβώς τι ρυθμίζουμε σήμερα, τι ρυθμίζουμε και θα συνεχίσει να ρυθμίζεται και στο μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε ακριβώς τι εννοούμε ρύθμιση των OTCs. Γιατί αυτό που σήμερα ρυθμίζουμε δεν σημαίνει ότι θα συμψηφιστεί και θα συνεχίσει να ρυθμίζεται και στο μέλλον. Καταλαβαίνετε ότι εκαθάριση, συμψηφισμός σημαίνει μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, συμπεριλαμβάνει το συστημικό κίνδυνο και μειώνοντας το σύστημα θα πρέπει να ξέρουμε αν ρουν οι νέες ρυθμίσεις το σύνολο αυτών των συναλλαγών, το σύνολο αυτών που σήμερα ονομάζουμε OTC. Κύριε Λάγκεν, είναι πολύ ενδιαφέρον να ξέρουμε αν αυτό που θεωρούμε ότι ρυθμίζουμε σήμερα θα το ρυθμίζουμε και στο μέλλον. Γι' αυτό και ήθελα να ξέρω για ποια παράγωγα ακριβώ μιλάμε. Η πρόεδρος έθιξε και ένα άλλο θέμα που με ανησυχεί. Τι ακριβώς ε, αναφέρουμε σήμερα στα χαρτοφυλάκια των ΟΤΙΣΗΣ. Ξέρετε πολύ καλά ότι όλος αυτός ο όγκος ε, συναλλαγών μπορεί από τη μία ώρα στην άλλη, από τη μία μέρα στην άλλη να μεταφερθούν και ένα τεράστιο τμήμα αυτών των συμβολέων και αυτών των συναλλαγών παραμένει σήμερα χωρίς ρύθμιση και θα ήθελα να είμαστε λίγο πιο προχωρημένοι στη ρυθμίσή μας. Σήμερα έχουμε μεγάλη καθυστέρηση. Βεβαίω δεν μπορεί κανείς σήμερα να υποχρεώσει όλους όσους έχουν αυτά τα προϊόντα στο χαρταφυλακιό τους να περάσουν από αυτό το clearing. Το backloading συνεχίζει να με απασχολεί. Ξέρω ότι ο κίνδυνος συνεχίζει να είναι τεράστιος. Και αυτό είναι μία από τις προσωπικές μου ανησυχία. Όσον αφορά την πρόσβαση στα δεδομένα, μιλήσαμε για διαλειτουργικότητα. Για μένα το καθοριστικό στο θέμα της διαλειτουργικότητας είναι τι απόφαση θα πάρουμε όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Θέλουμε ανταγωνιστικό περιβάλλον για τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους. Να έχουν δηλαδή όλη πρόσβαση στα ουσιαστικά δεδομένα. Από εκεί και πέρα να μπορούν να έχουν όλα τα στοιχεία και να μπορούν να περάσουν σε ένα συμπληφισμό. Τα δεδομένα και οι ροές των δεδομένων θα πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλους τους οργανισμούς συμψηφισμού. Εάν θέλουμε λοιπόν να έχουμε ανταγωνιστικό περιβάλλον, θα πρέπει αυτή η πρόσβαση να είναι εφικτή και πραγματική για όλους. Επίσης, δεν έχουμε συζητήσει ακόμα το θέμα των ε, συναλλαγματικών ισοτιμιών και αν αυτό θα είναι ή δεν θα είναι μέσα στο ρυθμιζόμενο περιβάλλον. Είναι η μεγαλύτερη αγορά, η αγορά spot για τις συναλλαγματικές ισοτιμίας θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην έκθεση αυτή. Αυτή είναι η δική μου άποψη και αν θέλουμε να ασχοληθούμε με την αγορά αυτή θα πρέπει να κοιτάξουμε όλες τις πτυχές γιατί και εδώ συμπεριλαμβάνονται τεράστιοι κίνδυνοι. Αν θέλετε η εκαθάριση είναι το πιο σημαντικό τμήμα αυτών των συναλλαγών και η αλλαγές ε, που θα, που θα επηρεάσουν τελικά αυτή την αγορά, είναι αλλαγές που θα πρέπει να τις αποφασίσουμε σήμερα. Και βεβαίως ο κίνδυνος που συμπεριλαμβάνεται εδώ είναι τεράστιος. Πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ο κύριος Λάγκεν βλέπω ότι είναι ανοιχτό σε κάθε συζήτηση και με μεγάλη ανεπομονησία περιμένουμε το κείμενό του. Πρόεδρος. Για τους συναδέλφους που μόλι μπήκαν, θα ήθελα να πω ότι ξεπεράσαμε λίγο το χρόνο για την έκθεση αυτή. Θα δώσω το λόγο ακόμα σε δύο μιλητές, ο κύριος Κλούτεν. schön. ich möchte... Ευχαριστώ πολύ. Ε, η προηγούμενη ομιλήτρια εκφράστηκε πολύ θετικά όσον αφορά τα παράγωγα. Εγώ εκ μέρου τη δική μου πολιτική ομάδα θα ήθελα να θέσω το γενικό ερώτημα κατά πόσο είναι αναγκαίο να βγει κανεί στην αγορά με τέτοιου είδου προϊόντα. Ε, πρόκειται για ένα ιδιαίτερο κερδοσκοπικό προϊόν και γενικά εμείς δεν βλέπουμε σε τι χρειάζεται κανείς τέτοιου είδους προϊόντα. Από την άλλη είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να το εξαφανίσουμε από προσώπου γης. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να κάνω αυτή την παρατήρηση. Θα ήθελα εν συντομία να πω κάποια πράγματα όσον αφορά τα τυποποιημένα και τα μη τυποποιημένα προϊόντα. Τα μη τυποποιημένα δεν είναι στην αρμοδιότητα των κεντρικών οργανισμών συμψηφισμού, γιατί δεν είναι διαπραγματεύσιμα δεν είναι δυνατόν μέσω ενός οργανισμού εκαθάρισης να εκαθαριστούν. Από την άλλη ανοίγεται με τον τρόπο αυτό η πόρτα σε μια υπονόμευση της συνολικής ε, ρύθμισης. Γι' αυτό θα έπρεπε να σκεφτούμε κατά πόσο δεν θα έπρεπε να συμπεριληφθούν ή να απαγορευθούν μάλλον και τα μη τυποποιημένα προϊόντα, να απαγορευθούν τα μη τυποποιημένα προϊόντα. Δεύτερον, σε σχέση με το θέμα των μη χρηματοοικονομικών αντισυμβαλόμενων. Θεωρούμε ότι έχει νόημα να μην το ορίσουμε ξεκάθαρα, ε, σε ποιο βαθμό δηλαδή ενέχουν σημαντικούς κινδύνους. Ε, όσον αφορά και μια τρίτη παρατήρηση, από τη δική μας σκοπιά δεν είναι αποδεκτό με τα να κάνει κανείς κερδοσκοπία με τα τρόφιμα και τις πρώτες ύλε. να κερδίσει κανείς χρήματα. Γι' αυτό θα θέλαμε ε, να απαγορευτεί αυτού του είδους το εμπόριο με τέτοιου είδους παράγωγα. Ο κύριος Λάγκελ είπε κάποια πράγματα σχέση με την εποπτεία και υπήρξαν κάποια σημεία τα οποία στηρίζουμε δηλαδή μια συνεπής εποπτεία όπω την παρουσίασε ο κ. Λάγκεν, υπό την προπόθεση ότι υπάρχουν τα προϊόντα αυτά, θα πρέπει να τα εποπτεύσουμε. Είναι ένα τρόπο να ρυθμίσουμε την αγορά. Αυτές ήταν οι παρατηρήσεις από τη δική μου σκοπιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η Βίκη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λάγκεν που ασχολήθηκε με τα εξαιρετικά πολύπλοκα θέματα. Όσον αφορά τη ε, σχέση με την ρευστότητα και τις ε, τράπεζες, το τραπεζικό σύστημα και την ε, MIFID, η οποία αναφέρθηκε εδώ. Θα ήθελα να θέσω το θέμα των εγγύσεων ρευστότητα για την υποστήριξη των κεντρικών αντισυμβαλόμενων. Από πού θα βρούμε αυτές τις εγγύσει, Όλα αυτά σχετίζονται με την κρίση βεβαίως του δημόσιου χρέους. Στην Επιτροπή Βασιλείας ορίζονται ε, ε, προβλέπεται ότι μέχρι το 2018 συγγνώμη, θα πρέπει να υπάρχουν νέοι κανόνες για τις ε, εγγύησεις. Ε, και βέβαια θα πρέπει να αλλάξει η φύση των επενδύσεων. Ένα άλλο πράγμα που συζητούμε είναι η συνεκτικότητα της νομοθεσίας, η απαιτούμενη συνεκτικότητα. Η Επιτροπή ε, μας λέει τα άπειρα τηλεφωνήματα που γίνονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα με ενδιέφερε να δούμε μία επιστολή που την Παρασκευή πήγε από το πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας ε, προς τον πρόεδρο της FTC ε, λέγοντας θα πρέπει να επιβραδυνθεί ο ρυθμός της θέσπισης των διατάξεων της νομοθεσίας γιατί θα πρέπει να υπάρξουν κανόνες, αλλά βεβαίως οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να είναι οι σωστοί. Ο κύριος Λάγκεν είπε επίση ότι θα πρέπει να έχουμε τους σωστούς ε, κανόνες και ε, θα πρέπει κάπως να επισπεύσουμε. Αλλά από την άλλη, εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται σε άλλες ε, περιοχές του κόσμου και θα πρέπει να γίνουν κάποιες μελέτες επιπτώσεων για να μπορέσουμε να κάνουμε μια εξολόγηση. Αυτό, εδώ έκλεισε ο κατάλογος των ομιλητών. Κύριε Λάγκεν, θέλετε να μιλήσετε. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα της ακρόασης του κυρίου Ντομινίτσι. Εδώ βεβαίως ε, δεν έχουμε κάποια ακρόαση. Θα πρέπει επίσης να τηρήσουμε τα χρονικά μας ε, περιθώρια. Βέρνερ, έχει λόγο ich bedanke mich. Ναι, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω. Θα είμαι σύντομο γιατί θα πρέπει να γίνει η ψηφοφορία. Ε, αφορά τι προτάσει, έχω σημειώσει όλε και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την πολύ πλατεία σα υποστήριξη. Θα ήθελα να τονίσω δύο θέματα, δύο σημεία. Όσον αφορά την ακρόαση, θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσο ή δυνατόν μεταξύ απόφασης στην Επιτροπή και Ολομέλειας να κάνουμε μία ακρόαση σε σχέση με τη χορήγηση εξαιρώσεων για το κατόφλι καθάρισης και επίσης για το θέμα των πρώτων υλών. Αυτό το δεύτερο θέμα, η αγορά των πρώτων υλών. Εδώ η Κομισιόν έχει υποβάλει μια δική της πρόταση, έχει εξαγγείλει μια δική της πρόταση, μια ανάλυση ε, όπου έχει, υπάρχει μια καθυστέρηση έπρεπε να γίνει αύριο. Ε, υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, θα την έχουμε όμως τις, επόλοιπες, ε, τις προσεχείς εβδομάδες. Ε, και θα έπρεπε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με αυτά τα τρία σημεία. Τώρα, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, εδώ υπάρχουν ορισμένοι υποστηρικτές της πρότασης της Ουγγρικής Προεδρίας και της πλειοψηφίας του Συμβουλίου. Θα πρέπει να γίνει σχετική συζήτηση. Νομίζω πρέπει να τηρήσουμε τις διεθνείς προδιαγραφές και τις δικές μας προτάσεις. Εάν δεν απατώμε, η Επιτροπή δεν θέλει να προχωρήσει αυτή την επέκταση σε όλα τα παράγωγα. Γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι σωστό ότι αν ρυθμίσουμε τα χρηματιστήρια θα πρέπει να υποβάλουμε μια ξεχωριστή πρόταση για αυτή τη ρύθμιση. Επίσης και το ζήτημα της κεφαλαϊκής επάρκειας θα πρέπει να συμπεριληφθεί εδώ. Ε, και εδώ υπάρχει ένας μηχανισμός πώς μπορούμε μέσω των κατεξοδότηση πράξεων να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε τις άλλες προτάσεις που ακόμα δεν έχουν τεθεί επιτάπητος. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει με την ε, MIFID και το CRD4. Ε, ο κύριος Κομφέ αναφέρθηκε σε ορισμένα σημεία τα οποία είναι αντικείμενα τροπολογιών, στα οποία δεν αναφέρθηκα, δηλαδή οι άδειες για τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους θα πρέπει να γίνονται από τις ε, χώρες εγκατάστασης, οι δε ε, άδειες για τα μικρόα, για τα αρχεία καταγραφής θα πρέπει να δίνονται από την ΕΣΜΑ μετά από ακρόαση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επεσήμενε ότι οι διεθνές ε, διαπραγματευθήσεις προδιαγραφές θα πρέπει να συμπεριληφθούν και όσον αφορά γέννη το θέμα των πρώτων υλών, συμμερίζομαι την άποψή σα, αλλά γέννη εγώ είμαι κατά των απαγορεύσεων. Τώρα, οι βραχυπρόθεσμε συναλλαγέ αφορούν μια άλλη έκθεση. Κατά πώ θα πρέπει να απαγορεύσουμε τι βραχυπρόθεσμε ε, κάλυπτε συναλλαγέ. Αλλά δεν είναι δυνατόν να ρυθμίσουμε την αγορά παραγόγων, συνάδελφε κύριε Κλούντεν, μέσω απαγορεύσεων. Εγώ είμαι υπέρ του να υπάρχει μια ε, διαφανής ε, ε ρύθμιση και βελτίωση που να μπορεί να καλύπτει τους ε, σημαντικούς ε, κινδύνους. Ευχαριστώ πολύ. Um, Ευχαριστώ. Νομίζω ότι τελειώσαμε με το σημείο αυτό. Προθεσμή για τις τροπολογίες είναι 15 Μαρτίου και θα τις εξετάσουμε στις 4 Απριλίου. Και τώρα θα πούμε ότι πρέπει να πάμε λίγο πίσω και να υιοθετήσουμε την ημερήσια διάταξη, κάτι που ξεχάσαμε να κάνουμε σήμερα το πρωί. Δεν αντιτίθεται κανείς, ωραία. Εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Και παρακαλώ πολύ όποιος εγκαταλείπει την αίθουσα να το κάνει με ηρεμία και ήσυχα. Η επόμενη συνεδρίασή μας με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανοικοδόμησης, του κύριο Τρισέ, την επόμενη εβδομάδα, στις 3. Στις 10 Φεβρουαρίου θα γίνει μια έκτακτη συνεδρίαση και στην ημερσία διάταξη έχουμε και την τροποποίηση της Ευρωπαϊκής συνθήκη. Σας παρακαλώ, μπορείτε να εγκαταλέψετε την αίθουσα ήρεμα, δεν χρειάζεται την ώρα που μιλάει η Πρόεδρος να μιλάτε, εάν θέλετε βεβαίως να επανέλθετε. Τέλος, μια έκτακτη συνεδρία θα λάβει χώρα και την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο, μάλλον μεταξύ 7 και 8.30 το βράδυ. Ζητώ συγγνώμη. Και επειδή κάλυψα τις, τα σημεία αυτά που έπρεπε να είχα καλύψει το πρωί, μπορούμε να περάσουμε στην έκθεση της κυρίας Ποδηματά. Α, όχι, συγγνώμη, έκανα λάθος. Υπάρχει ένα αίτημα του ΕΛΚ. 97, 94, 68 και 8. Οι τροπολογίες αυτές θα πρέπει να ψηφιστούν ξεχωριστά, είναι έτοιμα του ΕΛΚ. Μόλις μου το ε, έδωσε η γραμματεία, ελπίζω να μου το υπενθυμίσει. Τροπολογία 68. Η γραμματεία επιβεβαιώνει ότι η λέξη increased transparency, αυξημένη διαφάνεια, υπάρχει στο κείμενο της συμβαστικής τροπολογίας για την 97, 94 και 12. Η γραμματεία μου υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχει ασυμβατότητα με τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Εν πάση περιπτώσει, αν καταλαβαίνω καλά, καλύπτονται αυτές οι τροπολογίες από τις συμβιβαστικές. Η συμβαστική τροπολογία Β καλύπτει τις τροπολογίες αυτές. Αφού λοιπόν η συμβαστική τροπολογία Β ψηφιστεί, θα πάμε στην 15 και κατόπιν θα θεωρήσουμε εάν ψηφιστούν ότι οι συμβαστικές τροπολογίες αποτελούν το τελικό κείμενο. Κυρία Ποδηματά. Uh, uh, να σας ευχαριστώ. Θα ήθελα εδώ να πω ότι οι 94 και 97 τροπολογίες καλύπτονται από τις συμβεβαστικές. Και ιδιαίτερα η 94 καλύπτεται από το τελευταίο τμήμα της συμβαστικής H, ήτα, και το τελευταίο τμήμα της α. Και αυτό έχει συμφωνηθεί. Όσον αφορά την τροπολογία 97, πιστεύω ότι δεν είναι συμβατή αυτή η τροπολογία με την παράγραφο 8. Γι' αυτό και θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να ψηφιστεί ξεχωριστά. Ζων Πολ. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Σκιώδης. Τι έχετε να πείτε. Πολύ σύντομα, εχθές το βράδυ συμφωνήσαμε ότι αυτές οι δύο τροπολογίες δεν καλύπτονται. Δεν καλύπτονται. Γι' αυτό και το ΕΛΚ προτείνει αυτήν την ξεχωριστή τροπολογία. Όπως είπα, η γραμματεία συμφωνεί με την κυρία Χούντερ. Ζητώ συγγνώμη κυρία Πρόεδρε, αλλά εγώ είμαι πολύ καιρό σε αυτή την Επιτροπή. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι δεν είναι ευγενικό ένας κοιόδης εισηγητής να παρουσιάζει εδώ την άποψή του, η γραμματεία να συμφωνεί, αλλά η εισηγήτρια να μην έχει καν ρωτηθεί αν είναι συμβατό ή μη συμβατό το κείμενο. Αν διαβάσετε το κείμενο θα καταλάβετε ότι το περιεχόμενο δεν είναι συμβατό, δεν μπορεί να είναι συμβατό. Και ότι άλλο είναι το πνεύμα των συμβαστικών τροπολογιών. Γι' αυτό και θα σας παρακαλούσα σαν ε, πρόεδρο να παίξετε το ρόλο σας με ηρεμία και να μην ισχύσει εδώ άλλος κανόνας, διαφορετικός κανόνας. Ακολουθούμε την εισηγήτρια. Ναι, ναι. Την ακούσαμε όμως την άποψη της εισηγήτριας. Νόμιζα ότι οι <clears throat> πολιτικές ομάδες γνώριζαν και είναι πολύ δυσάρεστο το ότι οι συμβαστικές τροπολογίες εδώ δεν μπορούν να καλύψουν αυτά τα σημεία. Δεν μπορώ δυστυχώς να πάρω απόφαση χωρίς να κοιτάξω το κείμενο και να δω αν όντως καλύπτεται ή όχι. Μπορώ να δεχτώ όμως αυτό που λέτε ότι είναι άλλο το πνεύμα των συμβαστικών τροπολογιών. Τότε γιατί συζητάμε όμως. Με αυτή την έννοια καταλαβαίνω ότι θέλετε να παραμείνουμε στο κείμενο των συμβιβαστικών τροπολογιών, γιατί όλοι αυτό είχαν αρχικά προβλέψει και υπάρχει κατάλογος ψηφοφορίας και δεν μπορούμε να αποκλίνουμε από τον κατάλογο αυτό. Αν ε, δεν συμφωνούν οι πολιτικές ομάδες θα αναγκαστούμε να καταψηφίσουμε τις συμβιβαστικές τροπολογίες και να πάρουμε μία-μία τις τροπολογίες και να δούμε τι θα ψηφίσουμε. Μιλάμε για την 94, 97, 12. Κυρία Ποδηματά, για ποιες τροπολογίες ε, ζητούμε ξεχωριστή τροπολογία. 94-97 κυρίως. Και μπορούμε να ενημερώσουμε τα μέλη της Επιτροπής γιατί δεν είναι συμβατά τα κείμενα αυτών των τροπολογιών με τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Για να γίνει ξεχωριστή Μπορώ να σου το εξηγήσω. Όχι. Είναι το ίδιο Άρα θα παραμείνουμε στις συμβαστικές τροπολογίες. Ωραία. Σχέδιο συμβιβαστικής τροπολογίας Α. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Είναι πραγματική η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε πραγματικά. Έχουμε τρεις επιπλέον ΕΛΚ που ψηφίζουν. Ξέχασα την κάρτα μου. Ζητώ συγγνώμη. Ψήφισαν όλοι. Εγκρίνεται. Ωραία. Συμβιβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Το πρώτο τμήμα ψηφίζαμε. Το δεύτερο τμήμα τώρα του Β. Κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές Ελέγχουμε την 47. Ψήφισαν όλοι. Ωραία. Εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω το ίδιο εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική C υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Το αρχικό κείμενο. Το 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική δέλτα. D. Εγκρίνεται. 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ελέγχουμε. Την 58. Εγκρίνεται. 60. Πέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. πέντε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτή νομίζω. Αλλά ελέγχουμε. Ελέγχουμε. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίνεται. Δεν σηκώσετε όμως αρκετά τα χέρια σας. Ελέγχουμε την συμβαστική. Να σηκώνετε τα χέρια σας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ήτα H ξεχωριστή. Το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ζητάτε ξεχωριστή τροπολογία. Όχι. Ναι, ναι, παρακολουθώ. Η Άλντε ζητάει υπέρ αυτών των λέξεων κατά αποχές εγκρίνεται. Όχι. Ψηφίζουμε υπέρ των λέξεων αυτών. Or failing that. Εντάξει. Εγκρίνεται με μία ψηφοδιαφορά. Δεν έχω την κάρτα μου. Α, ναι. Το λέει και προσπαθούσα να καταλάβω τι μου έλεγε τόση ώρα. Ναι, αυτό είναι πρόβλημα. Είναι πολύ μικρή η διαφορά. Άρα καταπίπτει. Δεν εγκρίνεται. Έτσι. Ωραία. Προχωράμε στην συμβιβαστική γιώτα. Άι. Όχι. Υπέρ της γιώτα κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική. Μάλλον υπέρ κατά. Ποιος ψηφίζει. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 95 ψηφίζαμε την 8 καλύπτονται αυτές Α, τροπολογία 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική J τρία τμήματα ναι όχι Δεν είμαι σίγουρη ότι καταλαβαίνω, λέει η Πρόεδρος. Το πρώτο τμήμα είναι μέχρι τη λέξη market efficiency. Το δεύτερο είναι μέχρι το financial markets. Και το τρίτο τμήμα είναι ότι θα βγάλουμε μία μικρή φράση, το since και τα λοιπά. Ναι ή όχι, κατάλαβα καλά, λέει η πρόεδρος. Να μας εξηγήσει ίσως η συγγήτρια. Στην παράγραφο 9 υπάρχει μια προφορική τροπολογία των πρασίνων. Να αντικαταστήσουμε τη λέξη could με τη λέξη would. Το πρώτο που ψηφίζουμε. Και μετά μοιράζουμε την παράγραφο, όπως είπατε, μέχρι market efficiency και το δεύτερο από stresses μέχρι financial markets. Αλλά πρώτα έχουμε την προφορική τροπολογία των πρασίνων να βάλουμε τη λέξη good στη θέση της λέξης could. Ωραία. Οι πράσινοι ζήτησαν και μία άλλη ξεχωριστή ψηφοφορία. Since there is μέχρι το financial market. Ναι ή όχι. Το έχετε αποσύρει αυτό. Άρα, άρα κόφεται το τελευταίο τμήμα σε δύο. Αν δεν μου πείτε περί τίνος πρόκειται, δεν ψηφίζουμε. Ωραία. Κάνουμε αυτό που ζήτησε η εισηγήτρια τότε. Θα κάνουμε αυτό που είπε η συγγήτρια. Η προφορική τροπολογία των πρασίνων. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, ελέγχουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Δεν εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το τρίτο. Από το stresses μέχρι financial markets. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτό. Τέλος αυτής της ψηφοφορίας. Συμβαστική κάπα. Δύο τμήματα και εδώ. Το πρώτο από stresses μέχρι implement. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο από recalls μέχρι account υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται νομίζω και αυτό συμβιβαστική λάμδα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτό συμβιβαστική μη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται νη συμβαστική νη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική όμικρον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική π υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 126 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το συμβαστικό Q υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική ρο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική Σίγμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 141 δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο υπέρ κατά αποχές επίσης εγκρίνεται συμβιβαστική ταφ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γιου, συμβασική γιου, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβασική β, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και μετά 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ψηφίσαμε την 50. Ήταν τροπολογία Άλντε. Γιατί ανησυχεί εδώ η Άλντε. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 157. Ελέγχουμε. 157. Εγκρίνεται. 159 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει 61, 161. 162 εξήντα υπέρ. Όχι. Καταπίπτει. Ωραία. Καταπίπτει. Έτσι λέει η συγγετία. Συμβαστική W. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική X. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 168 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική ύψιλον. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 172 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 172. Εγκρίνεται. Ναι με μια ψηφοδιαφορά. 173 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε την 173. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Συμβιβαστική ζήτα. Υπέρ. Έχουμε τρία τμήματα. Το πρώτο. Υπέρ. Το πρώτο. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το δεύτερο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το τρίτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική αλφα. Το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ, κατά, αποχές, Τρία. Ένα. Αποχές. Ελέγχουμε. Να ψηφίσουν παρακαλώ πολύ όλοι. Ελέγχουμε. Καταπίπτει. Δύο, ήτρε δύο, υπέρ, κατά, ποχές, εγκρίνεται. Έξι, υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε. 6, ήτρε 6, ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίνεται. 9, 9, τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τρίτο, α, συγγνώμη, δέκα δέκα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έντεκα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. δώδεκα Το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Το δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε το 13 της Ήτρε. Καταπίπτει. 180 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 181 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 187 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Το αρχικό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 182 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 183 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 185 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 186 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΑΒ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 192 υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 192. Oh, some abstaining going on, so, right. everybody voted. Ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Ανάπτυξη 1 δεν ψηφίζεται. Δεν ανάπτυξη 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ήτρε 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ανάπτυξη 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ανάπτυξη 9 υπέρ, κατά, αποχές να ελέγξουμε την 9 της Επιτροπής Ανάπτυξης. So if okay. That's carried by one. Ψηφίσατε όλοι, εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Η επόμενη είναι η 17 ε, της Επιτροπής Ανάπτυξης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 193 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 194 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται νομίζω αλλά κάποιοι δεν ψηφίζουν, οπότε ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέντε, γιατί amendment yes. για την ψηφίζουμε, ε. εγκρίνεται. Συμβιβαστική AC υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AD υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΑΕ e, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AF υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AG υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. A υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AI υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AJ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33. Υπέρ κατά αποχές νομίζω πως απορρίπτεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αλλά ας ελέγξουμε, γιατί δεν είμαι σίγουρη, για την 34. Have Λοιπόν, εγκρίνεται όντως ε, η ένα υπέρ, μάλλον το αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, λέει η πρόεδρος. διαφωνείτε να το ελέγξουμε. Oh, a thumb's changed direction here. <laughs> yeah, okay. Uh, citation 2 to 6 in... Εκτιμώντας 1 μέχρι 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκτιμώντας 8 με 23 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Περιμένατε. Τι θέλετε. Ούντο. Κυρία Πρόεδρε, είχαμε μια ψηφοφορία που τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά από ό,τι είχε συζητηθεί μεταξύ των πολιτικών ομάδων και είχε συμφωνηθεί. Την περασμένη εβδομάδα είχε ζητηθεί μια εντελώ διαφορετική συμπεριφορά ψηφοφορία από αυτή που εκφράστηκε σήμερα. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που έπραξαν συνεπώς με αυτό το οποίο είχαν εκφράσει. Και είμαι κάπως εκνευρισμένος και απογοητευμένος με τη συμπεριφορά άλλων ε, παρακαλώ να κάνουμε μια διακοπή ενός λεπτού για να μπορέσουμε να συζητήσουμε εντός των πολιτικών ομάδων ούτε ώστε να αποφασίσουμε την οριστική ψηφοφορία, ε, την ε, συγγνώμη, συμπεριφορά κατά την ψηφοφορία. Όλε Σμιτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι εμείς ε, μείναμε πιστοί στις υποσχέσεις μας της προηγούμενης εβδομάδας. Anyway, um... Εν πάση περιπτώσει η σοσιαλιστική ομάδα ζήτησε ένα λεπτό να διαβουλευθεί γιατί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν ήταν το αναμενόμενο. Ενός λεπτού διάλειμμα πριν από την τελική ψηφοφορία. have we? I think. Udo, are we ready? Right, we'll take... Τι έγινε, Ούντα, είμαστε έτοιμοι. Να ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τι θες να πεις, Άννη, θες να πεις δύο λόγια. Thank you, Sharon. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σαν εισηγήτρια, θα ήθελα να προτείνω στους ε, συναδέλφους να ψηφίσουν υπέρ της έκθεσης μου, αλλά κρινά όμως πρέπει να σας πω ότι πιστεύω ότι μπορούσαμε να τα είχαμε πάει πολύ καλύτερα. Και όταν λέω ότι μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα διατηρούσαμε τις διαφορετικές μας προσεγγίσεις και θέσεις σε σχέση με κάποια θέματα κλειδιά, όπως π.χ. το EUFTT. Και κατά τη γνώμη μου αυτό που είναι ακόμα πιο σημαντικό από αυτό είναι να μπορούμε να υπερασπιστούμε την αξιοπιστία αυτού εδώ του σώματος και αυτής της Επιτροπής που είναι συνεπής με τα ε, κοινά το κοινό έδαφος το οποίο μπορέσαμε να βρούμε και να συνοηθούμε μετά από πολλές προσπάθειες και δυσκολίες. Ε, και πάλι να πω λοιπόν ότι πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει πολύ καλύτερα. Δεν είμαι 100% ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα, αλλά νομίζω πως έχουμε μερικές εβδομάδες μπροστά μας πριν την ψηφοφορία στην Ολομέλεια, ώστε να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που σου είπα μόλις, ότι δηλαδή να είμαστε πιο συνεπείς και συνεκτικοί με το κοινό τα κοινά στοιχεία στα οποία καταφέραμε να φτάσουμε μετά από πολλές προσπάθειες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. On the uh, text as Και ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Has Ψηφίσατε όλοι, τέλος της ψηφοφορίας. 30 υπέρ, 4 κατά και 6 εποχές.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 Έχουμε ακόμα ένα θέμα. Όσοι φεύγουν να το πράξουν εσύχω. Hmm. Edward, who is going first? Right, we're now moving on to agenda. Προχωράμε λοιπόν τώρα στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης, στην τροπολογία του άρθρου 136 της συνθήκης. Έχουμε δύο εισηγητές. Ποιο, ποιος θα μιλήσει πρώτος, ο Σικλούνα, ο Έντουαρτ. Ο Έντουαρτ Σικλούνα θα μιλήσει πρώτος. Thank you. Um, the background Ξέρετε ότι το, η βάση για αυτή την έκθεση είναι η απόφαση του Συμβουλίου που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω το ιστορικό γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι έκανε τα κρατημέλη στο Συμβούλιο να λάβουν την απόφαση που έλαβαν. Και επειδή είναι τέτοιο βήμα άνευ προηγουμένου, και η διαδικασία είναι αυτή που είναι, η ΑΦΚΟ, γνωμοδοτεί και εμείς το ίδιο γνωμοδοτούμε. Όσο γινόταν έχουμε κάνει διαβουλεύσεις μεταξύ μας, ώστε να ξετάσουμε ο καθένα διαφορετικό τομέα. Μα μας συνδέεται περισσότερο με του στόχους της Επιτροπής μας, ενώ η ΑΦΚΟ περιορίζεται σε θέματα διαδικαστικά. Ωστόσο, ορισμένε φορές υπάρχουν και επικαλύψεις. Και μπορεί κάποιοι συνάδελφοι να αναφερθούν σε αυτές τις επικαλύψεις στο μέλλον. Εγώ πιστεύω και εδώ συμφωνούμε με τις δύο οι δύο ομάδες που ανέλαβαν να εκπονήσουν αυτές τι γνωμοδοτήσει για το ότι ο μηχανισμός που προτείνεται είναι ένα απαραίτητο εργαλείο, ένα μέσο, όμως δεν είναι το μόνο, ο μόνος μηχανισμός, είναι ένας μηχανισμός μεταξύ άλλων και πρέπει να συνοδεύεται από άλλα μέτρα, πολλά άλλα μέτρα, που όπως ξέρουμε συζητώνται στην, στο πακέτο της για την οικονομική ε, διακυβέρνηση. Τα, στα εκτιμώντα στην ετυλική έκθεση καθιστούμε σαφή την έμφαση που δίνουμε στο συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή στην προσθήκη περαιτέρω συμπληρωματικών μέτρων παράλληλα με αυτό το μηχανισμό με στόχο τη μείωση των κινδύνων για την οικονομική σταθερότητα και την ενίσχυση των προληπτικών και διορθωτικών ε, μέτρων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Επίσης, επαναλαμβάνουμε ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη εποπτεία των, ε, της εκτέλεσης των προπολογισμών καθώς και νέε διαδικασίες σε σχέση με τις μακροοικονομικές διαφορές και αστάθειες. Το δεύτερο, στην δεύτερη λογική σκέψη λέμε ότι η αρχή της αλληλεγγύης ανάμεσα στα κάτι μελη της Ένωσης, ιδιαίτερα εκείνα που είναι μέσα στην Ευρωζώνη, είναι να αντιμετωπίσουν τα θέματα που είναι κοινά για την Ευρωζώνη, δηλαδή μέσω και μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα αλλά και αντιμετώπιση του θέματος των μακροοικονομικών διαφορών μεταξύ τους. Το άλλο θέμα αναφέρεται στο γεγονός ότι καθώς πρόκειται για μια συνθήκη, μια συγγνώμη, προσθήκη στη συνθήκη, δεν μπορεί να μπει στις λεπτομέρειες για όλα τα θέματα. Προφανώς θα υπάρξουν διαφωνίες, ορισμένοι αναφέρουν τα ευρωομόλογα, κάποιοι δεν είναι υπέρ και ούτω καθεξής, αλλά εμείς λέμε πως η Κομισιόν θα πρέπει να φτιάξει ένα λεπτομερή σύνολο κανόνων για το πώς θα διαχειρίζονται τους συγκεκριμένους κανόνες και έπειτα να διευκρινίσει ποια θα είναι τα άλλα μέσα μέσα στο πλαίσιο της εντολής της τέλος. Ε, όπως ξεκινήσαμε κιόλας, λέμε ότι η Κομισιόν θα πρέπει να εξετάσει και άλλους μηχανισμούς για να εξασφαλίσει την ε, δημοσιονομική σταθερότητα της Ευρωζώνης και να προβεί στις απαραίτητες νομοθετικές προτάσεις. Στρεφόμενοι τώρα στο ίδιο το άρθρο που προτείνεται από το Συμβούλιο, Εδώ πιστεύουμε ότι έχουμε κάπως σε διαφορετική εικόνα για αυτό το μηχανισμό. Εμείς θεωρούμε πως αυτός ο μηχανισμός, όποιος και αν τον διαχειρίζεται, θα δίνει τη δυνατότητα να συνεχίζουν οι εργασίες χωρίς αυτός να αποτελέσει ένα να είναι ένα μηχανισμός που πρέπει να ενεργοποιηθεί. Το να χρησιμοποιούμε λέξεις όπως η λέξη ενεργοποιώ σημαίνει πως είναι κάτι το οποίο ποτέ δεν εξετάζεται και που ε, βασικά πατάει κανείς ένα κουμπί τη στιγμή μόνο που το χρειάζεται. Ε, και ότι δεν πρόκειται για κάποιο μηχανισμό που λειτουργεί διαρκώς και κάνει κάποια συγκεκριμένη δουλειά. Και η άλλη λέξη που λέει ότι είναι απαραίτητο σημαίνει πως οι μάνατζερ του θα πρέπει να διαβουλεύονται και να προβαίνουν σε αυτό το πολύ σημαντικό βήμα ενεργοποίησης του μηχανισμού μόνο αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Δηλαδή, να είστε βέβαιοι πως το καράβι θα πουλιάξει 100% για να πατήσετε το κουμπί για να κατέβουν οι σωσίβιες λέμβοι. Εμείς πιστεύουμε λοιπόν πως η τροποποίηση της δεν χρειάζεται να γίνει με τόσο σημαντικές λέξεις και γι' αυτό νομίζω πως το άρθρο μπορεί να σταθεί και χωρίς αυτές τις λέξεις, να πούμε μόνο μηχανισμός διασφάλισης σταθερότητας. Και τώρα μετά με ποια μέσα θα, είναι, θα ακολουθεί. Αλλά εδώ πρόκειται για μια μόνιμη αλλαγή στη συνθήκη και δεν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τέτοιες περιοριστικές λέξεις που μπορεί να μας κάνουν τη ζωή πολύ δύσκολη στο μέλλον. Τώρα, ερχόμαστε στο τελευταίο, αλλά θεωρούμε πολύ σημαντικό στοιχείο, τη τελευταία προσθήκη. Θα θυμάστε ίσως και πολλοί το είπαν και ο Τρισέ και τότε βλέπουμε ότι ακόμα και ο Σόμπελ στις 26 Ιανουαρίου που έβγαλε λόγο είπε τα ίδια, είπε ότι βασικά δεν πρόκειται για κρίση του ευρώ, αλλά για κρίσεις σε μεμονωμένες χώρες του ευρώ τη Ευρωζώνη. Όταν μιλάμε λοιπόν για ένα μηχανισμό ή ένα ταμείο που θα βοηθήσει, θα βοηθήσει όχι άμεσα το ευρώ, αλλά θα, το κάνει, θα, θα, βοηθήσει τις μεμονωμένες χώρες που το χρειάζονται. Εμέσως θα βοηθήσει το ευρώ. Δεν μπορούμε λοιπόν να μην αναφερόμαστε στα μέλη της Ευρωζώνης. Από αυτά θα συμβάλλουν μέσα σε ένα πνεύμα αλληλεγγύης. Και αναμένουν να έχουν τη βοήθεια αν τη χρειαστούν. Πιστεύω και αυτή την πρόταση κάνουμε. Πως όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης θα πρέπει να ωφεληθούν από αυτό το μηχανισμό. Και να λέμε ότι αυτό θα χρησιμοποιείται ή θα ενεργοποιείται μόνο αν αυτό είναι απαραίτητο για να απειλείται στο σύνολό της η σταθερότητα της Ευρωζώνης στην ουσία επιβαρύνει κάθε χώρα ώστε να αποδείξει πως τα προβλήματά της, ε, το, το χρέος της και τα λοιπά και το, η κρίση στην οποία διανύει επηρεάζει το νευροζώνη γενικότερα. Πολλές χώρες μπορούν αυτό να το δείξουν χωρίς αμφιβολία, αλλά υπάρχουν μικρές χώρες που μπορεί να το βρουν δύσκολο να το κάνουν κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως όλοι οι, όσοι συμβάλλουν, ολόκληρη η οικογένεια της Ευρωζώνης θα πρέπει να μπορεί να ωφεληθεί από αυτόν τον μηχανισμό. και να αναφέρουμε ρητά ότι όλες οι χώρες μέλη της Ευρωζώνης θα μπορούν να ωφεληθούν από το μηχανισμό. Αυτές είναι συνοπτικά οι αλλαγές, οι τροπολογίες που προτείνουμε για αυτή με αυτή τη γνωμοδότηση. Φυσικά δεν αναφέρω τίποτα που έχει συζητηθεί με την ΑΦΚΟ για τις διαδικασίες για το που θα μπει δηλαδή το κάθε θέμα στην τάδε παράγραφο στη Δίνα, αυτό θα το αφήσω για την ΑΦΚΟ. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Ζαν Πόλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομα. Ε, θα πω ότι συμφωνώ με τις παρατηρήσεις του συνεισηγητού μου και θέλω να διευκρινίσω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι καταγοργώντας τη λέξη αναγκαίο θέλαμε να αποφύγουμε τη νομική συζήτηση. Γιατί όταν έχουμε σε ένα κείμενο κάποιες λέξεις που τελικά καταλήγουν σε μια εξολόγηση της κατάστασης, ε, διατρέχουμε τον κίνδυνο να εμπλακούμε σε μια τέρμονη συζήτηση για να διαπιστώσουμε κατά πόσο είναι αναγκαίο ή έχει, κατά πόσο αέρας που αναπνέουμε είναι αναγκαίος ή όχι. Ε, όταν είναι πολισμένος, ε, πάβει να είναι αναγκαίος ή όχι. Ωστόσο, ε, θέλαμε να έχουμε κάποιες αντικειμενικές διατάξεις, αυτό λοιπόν διαγράψαμε το αναγκαίο. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα της αλληλεγγύης με τις χώρες της Ευρωζώνης, θα έλεγα ότι η ρητή διατύπωση που διατηρήσαμε έχει σαν σκοπό να ανέξει τη συζήτηση, δηλαδή να μην αφήσει καμία αμφισημία εν σχέση με το, αυτό που αποκαλούμε οι δυσκολίες της Ευρωζώνης. Δηλαδή ή θεωρούμε ότι οι μηχανισμοί επίλυσης της κρίσης ή βοήθειας σε περίπτωση δυσκολίας του ευρώ είναι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά με έναν συνολικό τρόπο εάν το πρόβλημα είναι συνολικό για την Ευρωζώνη είτε όπως εξηγήθηκε υπάρχει μια δυνατότητα να παρέμβουν οι μηχανισμοί αυτοί αυτή στιγμή μία από τις χώρες της Ευρωζώνης έχει τέτοιες δυσκολίες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο να δημιουργήσουν πραγματικές δυσκολίες στην Ευρωζώνη. Εδώ λοιπόν προτείνω μια τροπολογία περισσότερο για να επιλέξουμε παρά να πούμε ότι αυτή είναι η εξεποκαλύψος ε, αλήθεια αυτής της τροπολογίας. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια, ένας βασικός προβληματισμός, δηλαδή ότι η τροποποίηση της συνθήκης και ας μην σκεφτούμε λοιπόν θα πρέπει να τροποποιήσουμε σβάθος το κείμενο, δεν θα πρέπει η τροποποίηση αυτή να δημιουργήσει νέες αμφισημίες. Κάνουμε νέες τροποποίησεις για να ικανοποιήσουμε ορισμένες θεσμικές απαιτήσεις ορισμένων ε, νομολογιών ορισμένων ε, χωρών δεν θα πρέπει, ορισμένων δικαιοδοτικών οργάνων ορισμένων χωρών, δεν θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε νέες αμφισημίες αυτή τη στιγμή σε εφαρμοστούν αυτοί οι μηχανισμοί. Ιδού λοιπόν και θα ήθελα να πω ότι υποστηρίζω τα όσα είπε ο προηγούμενος ομιλητής που είναι και ο συν Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους του Άλντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Συζητήθηκε το θέμα αυτό όταν άρχισε να ενισχύεται η ευρωπαϊκή οικονομία. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι όλα αυτά τα ευχάριστα δεν μπορούν να διαρκέσουν επάπειρον. Η κρίση μας έδειξε ότι πραγματικά είναι περίπλοκο το κοινό μας ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα και εμπεριέχει και κινδύνους για το μέλλον. Γι' αυτό και σε αυτή τη σημαντική στιγμή της ιστορίας μας. Χαίρομαι που έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν τα κρατημέλη ότι μπορεί να παραλύσει το σύστημα. Η Ευρωζώνη πρέπει να έχει μια προληπτική δράση έτσι ώστε να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και τα προβλήματα και να υπάρχουν κάποιες εγγύσεις για το μέλλον. Η Ευρωζώνη πρέπει να προστατευθεί και αν δεν είχε κάποια προστασία θα ήταν πολύ χειρότερη η οικονομική κρίση για κάποιες χώρες, μεταξύ των οποίων και η δική μου η Ισπανία. Θεωρώ ότι η πρόταση αυτή την οποία θα στηρίξω είναι ένα σημαντικό βήμα έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια καλύτερη οικονομική οργάνωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μια εγγύηση για καλύτερη σταθερότητα στο μέλλον. Τέλος, δεν πιστεύω ότι πρέπει να σταματήσουμε σε αυτό το διορθωτικό επίπεδο για να διασφαλίσουμε την σταθερότητα στην Ευρώπη χρειάζονται μηχανισμοί σταθεροποίησης για την πρόληψη κρίσεων και για την εξουδετερέση των επιπτώσεων της κρίσης. Θα υποβάλω λοιπόν και κάποιες τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, τι να προσθέσω. Καινούριο ή ήδη γνωστό που θα μπορούσε να προσθέσει κάτι σε αυτό το κείμενο. Η άποψή μου είναι ότι η διατύπωση σε αυτήν την αλλαγή που προτείνουμε έχει συζητηθεί ώρες ολόκληρες από τους επικεφαλείς κρατών μελών. Γι' αυτό και πραγματικά αναρωτιέμαι αν το οτιδήποτε προτείνουμε εδώ θα μπορούσε να περάσει από μια ψηφοφορία. Αν θα μας επιτραπεί δηλαδή κάτι να αλλάξουμε εδώ. σε αυτό το συμβαστικό κείμενο του Συμβουλίου. Η τροπολογία μου, την οποία έχω υποβάλει, οι τροπολογίες μου μάλλον, είναι τρεις. Αφορούν διατύπωση και κάποια αποσαφήνιση του κειμένου. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, η Σιλβή και άλλοι δύο μιλητές έχουν ζητήσει ο λόγο. Η Σιλβή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ τους εισηγητές. Εγώ θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση καταρχήν. Μετά από ε, το έντμα του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου μεταρρυθμίζουμε το κείμενο. Μήπως θα πρέπει να είμαστε όμως λίγο πιο απαιτητικοί και πραγματικά αυτό που εδώ με εκπλήσει είναι που η μεταρρύθμιση γίνεται μόνο στα αγγλικά και που τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι είναι τόσο επίγον αυτό το θέμα που δεν τηρείται η βασική αρχή της δημοκρατίας. Και το λέω αυτό και προς τον δικαστή, τον Γερμανό του Δικαστηρίου του Συνταγματικού της Καλτς Όσον αφορά το πακέτο για την οικονομική διακυβέρνηση, η κατάσταση είναι αρκετά περίπλοκη σήμερα. Αρχικά μας είπαν ότι δεν μπορούμε να ξανανοίξουμε τις συνθήκες. Η Επιτροπή λοιπόν πέρσι το καλοκαίρι υπέβαλε μια σειρά μέτρων προς τη σωστή κατεύθυνση, λέγοντας ότι δεν θα ακουμπήσουμε το κείμενο των συνθήκων. Τρεις μήνες αργότερα βλέπουμε, και θα το πω στον συνάδελφο ότι όντως τα κοινοβούλια κάτι θα πρέπει να χρησιμεύουν. Ναι, σκεφτήκανε οι επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων, αλλά υπάρχει και ένας κοινοβουλευτικός έλεγχος. Ναι, μπορούμε λοιπόν από ό,τι μας λένε σήμερα να ξαναδούμε το θέμα, να ξανανοίξουμε τη συζήτηση και μιλάμε για ακριβώς αυτό το συγκεκριμένο θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης. Ενίσχυση των κυρώσεων, οι μη αυτόματες τόματες κυρώσεις, δεν ξέρω ακριβώς, και κατά κάποιο τρόπο ξεπερνάμε το άρθρο 126 της συνθήκης. Εγώ λοιπόν προσωπικά θα κάνω προτάσεις, μπορεί να απορριφθούν αυτές, αλλά θεωρώ ότι αν το 136, το άρθρο 136 που αφορά τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν στη ζώνη ευρώ, πρέπει να δείξουμε συνοχή. Τα μέτρα της οικονομικής διακυβέρνησης θα πρέπει να είναι συνεκτικά και να μην μπορεί να υπάρξει καμία αμφισβήτηση. Σας ζητώ λοιπόν να μην δέχεσαι αυτές τις εξαιρετικές διαδικασίες, τις εντολές του Συμβουλίου, γιατί από ό,τι φαίνεται αποφασίζουν και διατάσσουν. Διαφωνώ. Δεν μπορεί επειδή αποφασίζει το Συμβούλιο το Κοινοβούλιο να εκτελεί. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είχα τελευταία ότι η πολιτική μου ομάδα το βλέπει με πολύ κριτικό βλέμμα. Όχι ότι είμαστε κατά κάποιων αλλαγών, αλλά θεωρούμε ότι αυτή την επισφασμένη διαδικασία θεωρούμε ότι δεν είναι εντάξει. Ε, Παρ' όλα δεν μπορούμε τώρα να την αλλάξουμε, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι εδώ διαπιστώνουμε ένα δημοκρατικό έλλειμμα, δηλαδή ότι γίνεται μια αλλαγή με μια τέτοια ταχύτητα. Επίσης δεν είμαι βέβαιος όταν βλέπω το ισχύον κείμενο κατά πόσο είναι αναγκαίο, απολύτως αναγκαίο να αλλάξει. Δηλαδή μπορούμε να διαβάσουμε το ισχύον άρθρο 136 λέγοντας ότι καλύπτεται η λεγόμενη οικονομική διακυβέρνηση. Τουλάχιστον αυτό δεν το αποκλεί η γερμανική μετάφραση, έτσι όπως εγώ τη διαβάζω και την κατανοώ. Δεν ξέρω λοιπόν, δεν είμαι απολύτως βέβαιος κατά πόσο είναι αναγκαία η αλλαγή. Και αυτό το οποίο έχω μπροστά μου στα αγγλικά όσον αφορά την ε, αλλαγή, την τροποποίηση, θεωρώ ε, της διατύπωσης strict conditionality, δηλαδή την, ε, την επιβολή αυστηρών όρων, θεωρώ ότι δεν είναι ενδεδειγμένη. Ε, αν από τη γερμανική οπτική γωνία αυτό θα μπορούσε να εισαδυναμεί με κάποιο είδου αυτοματισμό εδώ όσον αφορά τους όρους αυτούς. Κατά τα άλλα, σε σχέση με τις προτάσεις που έγιναν από τους οσηγητές, ε, θεωρώ ότι ε, μπορούμε να στηρίξουμε εδώ. Γιατί έχει νόημα να θέσουμε το ζήτημα της αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών μελών. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια σωστή πρωτοβουλία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μέντες Στεβίγκο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα το πρωί η Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων είχε μία συζήτηση σε σχέση με τη νομική εμβέλεια της αναθεώρησης, την οποία δεν πρόκειται εδώ να επαναλάβω εδώ. Αλλά θα ήθελα να εκφράσω μία σκέψη σε σχέση με το οικονομικό υπόβαθρο της, του ζητήματος. Εγώ συμφωνώ με τα όσα είπε ο εισηγητής ε, λέγοντας ότι η διαφορά μεταξύ αυτού το οποίο προτείνεται στο κείμενο του Συμβουλίου Δηλαδή αυτός ο μηχανισμός διαφύλαξης, δεν είναι ο μηχανισμός διαφύλαξη, αλλά είναι ένας από τους μηχανισμούς, ένα από τα τμήματα εδώ. Δεν θα πρέπει αυτός ο μηχανισμός να ισοδυναμεί με το γενικό πλαίσιο της λεγόμενης οικονομικής διακυβέρνησης, όπου υπάρχουν διάφορα τμήματα τα οποία εξετάζει αυτή η Επιτροπή από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο μέχρι τις έξι, έξι νομοθετικά τμήματα ή το ζήτημα των ευρωομολόγων και την πολεμική σχετά, σχετικά με τα ευρωομόλογα κλπ. Νομίζω ότι θα διαπράττουμε ένα σφάλμα αν θέλαμε να μετατρέψουμε αυτό το στοιχείο σε κάτι τόσο ουσιώδες. Τι θέλω να πω με αυτό. Εάν αποφασίσουμε ότι θέλουμε να μετατρέψουμε αυτό το κομμάτι σε ένα θεμελιώδες εργαλείο της Ευρωζώνης, νομίζω ότι θα μειώσουμε την προσοχή μας προς τα άλλα εργαλεία. Συνεπώς, όσον αφορά την ουσία και τις προταθήσεις τροπολογίες, με ανησυχεί η μνήα που έκαναν οι συγητές, όχι όσον αφορά τη συμπερίληψη των χωρών μελών γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτό το οποίο προτείνεται εδώ, αυτό το οποίο προτείνουν οι εισηγητές, ε, ε, αποκλεί ε, ε, είναι ε, ισοδομή μάλλον συγγνώμη, με ένα σχέδιο διάσωση για τι χώρε που αντιμετωπίζουν οικονομικέ δυσχέρειες. Και θεωρώ ότι αυτή δεν είναι η, η πρόθεσή μα. Εδώ αναφέρεται και είναι αλήθεια ότι πρόκειται για μια συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου. Αλλά το Συμβούλιο θα αποφασίσει εν σχέση ε, με αυτό και ποιο είναι το δικό μας περιθώριο λιμών, ε, δεν ξέρω, είναι περιορισμένο. Ωστόσο θα έπρεπε να γίνει μια σοβαρή προσπάθεια προβληματισμού εν σχέση με το αν επιβαρύνουμε πάρα πολύ το Ταμείο Σταθερότητας τελικά δεν μειώνουμε την εμβέλεια των άλλων εργαλείων τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας εντός ε, των άλλων νομοθετικών ε, τμήματων. Κύριε Πρόεδρε, εγώ πρόκειται να υποβάλω κάποιες τροπολογίες υπό την έννοια του περιορισμού της εμβέλειας του Ταμείου Σταθερότητας ούτω ώστε να μην συμπεριληφθούν σε αντίθεση ε, με την ε, πρόταση των εισηγητών ή χώρες μέλη. Θα παρουσιάσω τις ε, τροπολογίες αυτές, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ θέλω να πω δύο λόγια. Εγώ είμαι μεταξύ εκείνων που υποστηρίζουν ότι δεν χρειάζεται να αλλάξει η συνθήκη για να εισαχθούν ε, του είδους οι μηχανισμοί που έχουμε εισάγει. Και γι' αυτό φοβούμε ότι αν δεν έχουμε ακριβείς τροπολογίες, κλείνουμε μια πόρτα που παλιότερα ήταν, που ήταν ανοιχτή. Και νομίζω πως ο Έντουαρτ μας έδειξε πώς μπορεί να κλείσουν οι πόρτες για ένα κράτος μέλος που είναι μικρό και που η κατάρρευση του ποτέ δεν θα επηρέαζε την ε, σταθερότητα της Ευρωζώνης. Και εκτιμώ τις προσπάθειες που έχει καταβάλει. Κατανοώ το πρόβλημα της επιλογής των συγκεκριμένων λέξεων. Θα το σκεφτώ Μήπως ε, έχω καμιά φαϊνή που μπορεί να σημαίνει τα ίδια αλλά με διαφορετικά λόγια και ο κύριος Μέντες Δεβίγκο μπορεί να το καταφέρει αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει υποστηρίζω τις αλλαγές και να πω ότι πιστεύω πως η αρχική διατύπωση που προτάθηκε και συζητήθηκε από τα κράτη-μέλη θεωρώ πως είναι αρκετά επικίνδυνη. Και δεν βοηθάει και σε τίποτα. Μακάρι το Συμβούλιο να ακούγε λίγο περισσότερο τα όσα λέει το Κοινοβούλιο μας. Γιατί με το πέρασμα του χρόνου συχνά φαίνεται να έχουμε πιο πολλές φορές δίκιο από ότι το Συμβούλιο. Τώρα, έχουμε προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 3 Φεβρουαρίου το μεσημέρι. Δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Και έπειτα η εξέταση των τροπολογιών προβλέπεται για τις 10 Φεβρουαρίου. Ψηφίζουμε στην Επιτροπή στις 14 Φεβρουαρίου, στο Στρασβούργο δηλαδή τη Δευτέρα και η ψηφοφορία στην Αύκο στις 17 Φεβρουαρίου ώστε να μπορέσουμε να το περάσουμε από την πρώτη ολομέλεια του Μαρτίου, αν μπορέσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Φοβούμαι, όπως ήδη τονίστηκε, πως ε, φαίνεται πως θα δουλέψουμε στα αγγλικά. Δεν έχουμε τίποτα στα διάφορα για την επίσημη συνεδρίαση της ε, Επιτροπής μας. Επόμενη μας συνεδρίαση είναι Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου και τώρα έχουμε μία κυκλισμένο το θυρών συζήτηση σε σχέση με τους εκτελεστικούς ε, διευθυντές των διαφόρων αρχών. Όσοι συμμετείχαν σε εκείνη τη συζήτηση μπορούν να φύγουν, οι υπόλοιποι καλούνται να αποχωρήσουν.